How are you? Oh, <laughs> Having a great week? Yeah. <laughs> Colleagues, good morning. Can we reconvene the... Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. ξεκινώντας από τις ανακοινώσεις του Προέδρου θα αναφερθώ στη συνεδρίαση των συντονιστών τη χθεσινή. Όσον αφορά τον ορισμό εισηγητών και συντακτών, είχαμε έκθεση περιστατιστικών στοιχείων για τον τουρισμό. Καμία πολιτική ομάδα την ήθελε, οπότε είναι στα χέρια του Προέδρου οι συντονιστές αποφάσισαν για τη σύσταση, για την γνωμοδότηση για τους κανόνες και γενικές αρχές σχετικά με μηχανισμούς για τον έλεγχο από κράτη-μέλη των εφαρμοστικών εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια της γνωμοδοτήσεις που έχει το πιο σύντομο τίτλο στην ιστορία. Αντιθέτως, αστείευομαι. Είναι τίτλος «Σιδηρόδρομος». Είναι απλώς θέμα συναπόφασης. Η άποψη των συντονιστών είναι ότι ο εισηγητής θα έπρεπε να είναι από τις δύο, τους δύο μόνιμους εισηγητές που ασχολούνται με τη διαδικασία επιτροπολογίας και ο κ. Κούν που είναι ένας από αυτούς είναι ήδη εισηγητής για μία από τις άλλες επιτροπές και γι' αυτό αποφασίσαμε να δώσουμε στον άλλο εισηγητή της Επιτροπολογίας, τον κύριο Αλκατράουι, το θέμα για το προσθετικό ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συνέπειες της θέσης ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας για τις διάφορες διαδικασίες δημιουργίας θεσμών. Οι συντονιστές έλαβαν το φυλάδιο σχετικά με την Επιτροπολογία, το newsletter, είναι απλώς προς ενημέρωσή σας. Ε, είχαμε πολλά διάφορα. Τέθη διαδικαστικό. Το έθεσα ο υποφαινόμενος όσον αφορά στατιστικά στοιχεία για τη μεταφορά αγαθών και επιβατών δια της θαλασσίας οδού. Αυτή είναι η έκθεσή μου. Ενημέρωσα τους συντονιστές λέγοντας ότι η Ισπανική Προεδρία ήθελε να υιοθετηθεί αυτή η έκθεση κατά τη διάρκεια της Προεδρίας αυτής. Αυτό θα σήμαινε την εφαρμογή της απλουστευμένης διαδικασίας και την χρήση της αγγλικής γλώσσας ως γλώσσας εργασίας. Οι συντονιστές συμφώνησαν να ακολουθήσουν τις συνήθεις διαδικασίας, δηλαδή σχέδιο εκθέσεως για την Επιτροπή Μεταφορών, που θα συζητήσει στην Επιτροπή τέλος Μαΐου ψηφοφορία στη συνεδρίαση 21η 22 ιουνιου και μετά ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον μήνα Σεπτέμβριο η συζήτηση για τον μαύρο κατάλογο των, εταιριών, των αεροπορικών εταιριών αποφάσισαμε να μην συνεχιστεί συζήτηση και το ψήφισμα θα παραμείνει στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη στις 19 Απριλίου. Όσον αφορά τη συνέχεια που θα δοθεί για τις διακοπές και την αταναχή στις αερομεταφορές στην Ευρώπη, κατόπιν πρωτοβουλία του κυρίου Γκρός, του συντονιστού του ΕΛΚ και μετά από διεξοδική συζήτηση των συντονιστών απεφασίστη να υποβληθεί προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εις Ολομέλειων εκ μέρους της Επιτροπής Μεταφορών σχετικά με τις συνέπειες των διαταραχών των αερομεταφορών στην Ευρώπη, εστιαζόμενοι όλο ιδιαίτερο επί των δικαιωμάτων των επιβατών, το θέμα των αποζημιώσεων για τον τομέα των αερομεταφορών και την ανάγκη προώθηση ταχύτερη συντονισμένη εφαρμογή της νομοθεσίας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό με τη δημιουργία διαφόρων τμήματων, πλότ, λειτουργικών τμήματων τεναρίου χώρου και θα έπρεπε να προετοιμαστούμε και για τις 4 Μαΐου που θα γίνει το Συμβούλιο ε, Μεταφορών και το συζητούμε με τους συντονιστές και επεξεργαστούμε προφορική ερώτηση βάσει της πρωτοβουλίας του κυρίου Γκρός για τη Συμφωνία Αερομεταφορών Ευρωπαϊκής των τη Αμερική, οι συντονιστές, αποφ... αποφάσισαν να συμφωνήσουμε δική μου πρόταση, να ζητήσουμε από τον Επίτροπο, τον κύριο Κάλλα, να προβεί σε δήλωση στην Ολομέλεια όσον αφορά το θέμα αυτό, τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ενώση Αμερική και θα ακολουθήσει ένα ψήφισμα. Και αυτό θα πρέπει να προγραμματιστεί εγκαίρω πριν υιοθετηθεί η Συμφωνία από το Συμβούλιο Μεταφορών τέλο Ιουνίου. Υπάρχουν διάφορε επιλογέ που είχαμε σχετικά με το θέμα αυτό. Όμως η ταχύτερη λύση και που εξασφαλίζει ότι η γνωμοδότησή μας υποβάλλεται πριν από το Συμβούλιο ή εκφράζουμε τις σκέψεις μας πριν από το Συμβούλιο να εκφράσει τη θέση του, είναι η λύση να ζητήσουμε τον Επίτροπο προβεί σε δήλωση, διότι τότε δεν έχουμε τη φασαρία να προσπαθήσουμε να βρούμε χρόνο στην Ολομέλεια για, τα, για τις άλλες μεθόδους που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε. Επίσης υπήρξε πρόταση της ομάδας των Πρασίνων, του κυρίου Κράμερ, να συζητηθεί το ατύχημα που δημιουργήθηκε από ελκυστήρα γεωργικό εις Βέλγιον, όπου αρκετοί ποδηλάτες απόλυσαν την ζωή τους. Και σχετικά με αυτό ε, οι συντονιστές ε, συμφώνησαν με την πρόταση του Προέδρου ήτι; ότι θα πρέπει να συναντηθούν και να υποβάλουν προτάσεις για την επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών σχετικά με την αντιμετώπιση του θέματος εν τη ευρυτέρα ενία του όρου, όχι απλώς να περιοριστούν σε ένα και μοναδικό κράτος μέλος. Αυτά λοιπόν, σχετικά με τα όσα είπαν οι συντονιστές. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε εχθές. Έχετε σχόλια σχετικά με το θέμα. Η κυρία Φωστά έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, ναι, ένα σύντομο σχόλιο. Μας ειδοποίησαν σχετικά με το θέμα. Ζητήθηκε να έρθει κάποιο από την ΙΑΣΑ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφαλεία, να παραστεί στην συνεδρίαση Επιτροπή Μεταφορών στο μέλλον, διότι υπάρχουν ανησυχίε παντού όσον αφορά τη διαμόρφωση κανόνων και κυρίω σχετικά με τη χρηματοδότηση. Οπότε απογοητευθήκαμε τα μάλα, διότι αυτό δεν υποστηρίχθηκε από τι άλλε ομάδε, τι άλλε πολιτικέ ομάδε που είναι στην Επιτροπή. Υπάρχει άλλο άλλα σχόλια. Καλώ. Δεχόσαστε δηλαδή. Ε. Η κυρία Αγιάλα. Ετοιμάζουμε. Εφόσον ετοιμάσουμε την ερώτηση για το έγγραφο της Επιτροπής, ίσως θα μπορούσαμε να φροντίσουμε και για μια μικρή ακρόαση. Και να καλέσουμε, εννοείται και την ΙΑΤΕ και όλες τις οργανώσεις που έχουν εμπλεχθεί για να ακούσουμε και την δικιά τους άποψη. Αν πήγε περισσότερο, δεν ξέρω. Για σκεφτείτε το. Σας ευχαριστώ. Τώρα είμαι στα χέρια των συντονιστών σχετικά με αυτό το θέμα όταν θα καταλήξουν σε κάποια διατύπωση. Αν αυτή είναι μία από τι επιλογέ που θέλουν να εξετάσουν, αυτό αυτού αφορά. Σίγουρα δεν προτάθηκε αυτό μόνο σήμερα. Το αφήνω σε εσά αν θέλετε να κάνετε αυτή την πρόταση. Ωραία. Άλλο για τους συντονιστέ. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να πείτε, θεωρώ ότι συμφωνείτε. Ο κύριο Ντιγκράντε Πασκάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι για τον τουρισμό θα μιλήσει ο πρόεδρος της Επιτροπής. Ξανά την ερώτηση. Ναι, πρόεδρε, λέω. Για τον τουρισμό. Ο πρόεδρος της Επιτροπής θα τον αναλάβει. The tourism statistics. Yes, Για τα στατιστικά του τουρισμού. Αλήθεια, ναι. Δεν το ήθελε καμιά ομάδα και τον έλαβε ο πρόεδρος, εντάξει. Συμφωνούμε. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Πάμε παρακάτω. Επόμενο σημείο. Τους κοινωνικούς κανόνες για τον τομέα των οδικών μεταφορών. Η κυρία Ράμ έχει κάνει την έκθεση. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, Έχετε όλοι τις κάρτες ψηφοφοριών, θα γίνει δοκιμή τώρα. Δοκιμή, δοκιμή πρώτα, δοκιμαστική ψηφοφορία. Κύριε Κάντσιν, εγώ δεν έχω την κάρτα, δεν την έχω. Θα ψηφίσω με το χέρι λοιπόν, σκόντω το χέρι, για το πρώτο τμήμα. Εντάξει, δεν έχετε κάρτα, από ό,τι κατάλαβα. Έχετε όλοι τις κάρτες ψηφοφοριών. Ωραία. Μάτιο. Λοιπόν, να, να, να, να. Δυστυχώς η κάρτα Visa δεν μέτρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν περνάει. Ωραία. Να κάνουμε μια δοκιμή λοιπόν. Και ο κύριος Γκρός θα σηκώσει το δάχτυλό του, ξέρω εγώ τι άλλο θέλει. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Χώστε το, χώστε το. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν όλα τα δάχτυλα συντονισμένα με τον εγκέφαλο. Πέρας ψηφοφορίας. Ωραία. Εντάξει, υπέρ της δοκιμαστικής ψηφοφορίας είναι το αποτέλεσμα. Ξεκινάμε με την παράγραφο 1. Τροπολογία 6 του κυρίου Μπαχ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το 8 Lightfried. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 21 κατά. Διότι δεν έχουν δύο μέλη την κάρτα ψηφοφορία, και αυτό σα αναφέρω. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. 9, 9, 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές έλεγχος της τροπολογίας 10 του κυρίου Trade. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 25 ψήφοι κατά. Απορρίπτεται. 11 Free υπέρ. Κατά αποχές θα γίνει έλεγχος. Υπάρχει μικρή διαφορά σχέση με το παρελθόν. 11 ξεκινά ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες πέρα ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 21 κατά, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά σε ελέγξουμε. 12. Άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 20 υπέρ, 21 κατά, απορρίπτεται. 13 Bradburn υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται α, συγγνώμη, απορρίπτεται 17 α, απορρίφθηκε 16 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην παράγραφο 9. Κατά τμήματα ψηφοφορία ζητήθηκε από την ομάδα ECR. Πρώτα τονίζει ότι μέχρι σε όλα τα κράτη-μέλη και το δεύτερο καλεί τα κράτη-μέλη και το καθεξής. Πρώτο τμήμα. Περ κατά αποχές εγκρίνεται Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 Votman Call, προφορική τροπολογία που έχετε στα έγγραφά σας μπροστά σας υπέρ της προφορικής τροπολογίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Μετά πάμε στην παράγραφο 10, συμβιβαστική τροπολογία 1. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη είναι 21 του κ. Βαντάλεν υπέρ. Κατά 21, 21 δίκαιο έχει. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 25 είναι η επόμενη της κυρία Τσικάου. Υπέρ. Κατά. Αποχές θα κάνουμε έλεγχο, διότι τα χέρια πηγαίναν από εδώ και από εκεί. 25 της κυρίας Τσικάου ε, ξεκινά ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. 26 του κυρίου Μπράντμπερν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 Αγιάλα Σέντερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 Bradburn υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 γλωσσική αλλαγή, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 απεσύρθη, 32 ε, υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 33 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 34 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 35 με προφορική τροπολογία του κυρίου Ρικέ το έχετε, το κείμενο, η προφορική τροπολογία υπέρ, με την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 που αφορά την παράγραφο 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα πιο κάτω στη 46, όλες οι άλλες καταπίπτουν, μέχρι τη 46 καταπίπτουν. Ντανέλης, 46, 46, 46, έξι, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 43 του κυρίου Ελ Καντράουι. Την ψηφίζουμε σαν νέα παράγραφο. Έχουμε νέα παράγραφο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 του κυρίου Μπράντμπερν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ Μόνο η 47 εγκρίθη, αν εγκρινόταν η 47 περίφθη. Λοιπόν 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά πάμε στην 54. Και έχετε και προφορική τροπολογία στον κατάλογο ψηφοφορία της κυρίας Τικάου 54 με την προφορική τροπολογία. Αφορά την παράγραφο 18.1.9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 του κυρίου Κοχ, ξανά με προφορική τροπολογία της ηγήτριας, αντικαθιστά το, συ, το φορέα συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 55 με την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 57, συγγνώμη, Παράγραφος 19α, κυρία Τσικάμου, προφορική τροπολογία, υπέρ λοιπόν, 57 υπέρ. Το ΕΛΚ είναι κατά από ό,τι καταλαβαίνω. Αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 της κυρίας Λίχτεμπεργκερ. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπογραμμίζει μέχρι από, την, από τις ελέγχουσες αρχές, δεύτερον παροτρύνει κλπ. κλπ. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, θα γίνει έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας κάνουμε έλεγχο. Για το δεύτερο τμήμα της 59 ξεκινά ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Πράγματι, πράγματι απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Παράγραφος 20. Α, συγγνώμη. 60 Βαντάλεν. Για την παράγραφο 19α, 9. 60 Βαντάλεν υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος για την 60 Βαντάλεν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 22-19 ψήφους. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 οι 62 και 64 αποσύρθηκαν. Οπότε πάμε στην 61. Κοχ. Υπέρ. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, γκρίνεται. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67. Απεσύρθη. 68. Ε, υπάρχει κατά τμήματα ψηφορία που ζήτησε η ΑΛΤΕ. Πρώτο τμήμα. Με προφορική τροπολογία του κυρίου Αλκαντράουι. Θεωρεί ότι διαθέσιμη τεχνολογία και όλο αυτό το κείμενο, μέχρι εκεί που λέει κράτη-μέλη, συμπεριλαμβάνοντα όμω την προφορική τροπολογία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από γειτονικέ χώρε και το δεύτερο τμήμα είναι τα υπόλοιπα. Είναι ξεκάθαρο τι ψηφίζουμε. Πρώτο τμήμα τη 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές και το δεύτερο τμήμα και αυτό εγκρίνεται. 69 της κυρίας Λίχτεμπεργκερ υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 21, συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 3, υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Οπότε 71 έως 74 καταπίπτουν, η 70 απεσύρθη, οπότε πάμε στην 75. Έχω αρχίσει να μαθαίνω. Κατά τμήματα ψηφοφορία για την τροπολογία του κ. Μπράτμαν, πρώτα απ' όλα έχουμε τη διαγραφή των λέξεων και ούτω ώστε να διεξάγονται έλεγχοι αποτελεσματικά, να διαγραφεί αυτό. Και το δεύτερο τμήμα είναι η λέξη ασφάλεια. Λοιπόν, το πρώτο τμήμα Τις 75 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές Μπορούμε να ελέγξουμε την 76 σας παρακαλώ Τη Ξεκινά ο ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι σας. Τέλος ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις πάμε. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2, υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. τρία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. πέντε απεσύρθη. Τελική ψηφοφορία η οποία ξεκινάει. Ψήφισαν όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 35, 37 υπέρ, 5 κατά, 37 υπέρ, 5 κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν, κυρία Ράνερ. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η διεύρυνση και πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ντεβιράκ. Δύο λεπτά, Κριστίν, μέχρι να αποχωρήσουν ησύχω από την αίθουσα όσοι θέλουν να αποχωρήσουν. So if you're leaving, can you please Όσοι αποχωρείτε, παρακαλώ, ησύχω αν πάλι παραμένετε στην αίθουσα και πάλι ησύχως να παραμείνετε, ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε την εισηγήτρια. Okay. Καλώς. Παρακαλώ, κύριε Ντεβεράκ, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην παρουσίαση αρχές Μαρτίου του εγγράφου εργασίας μου, με στηρίξατε όσον αφορά τις προτεραιότητες που εντόπισα τότε. Ακολούθησα λοιπόν αυτή τη γραμμή και έτσι οι περισσότερες τροπολογίες έχουν να κάνουν με τους δύο κύριους στόχους πάνω στους οποίους συμφωνήσαμε. Δηλαδή να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των ερευνών όσον αφορά τα αεροπορικά ατυχήματα μέσω δικτύου και να ενισχύσουμε τη στήριξη στα θύματα και τις οικογένειές τους. Όσον αφορά καταρχήν τα δίκτυα. Μια στιγμή, Κριστίν, μια στιγμή να σε διακόψω, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν προβλήματα με κάποια γλώσσα διερμηνίας. Τα ελληνικά ακούγονται καλά, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τα δίκτυα που είναι υπεύθυνα για τις έρευνες και την ασφάλεια. Υπάρχουν τα εθνικά γραφεία διερεύνησης που ασχολούνται με τις περιπτώσεις ατυχημάτων. Η ποιότητα της εργασίας είναι αυτή η οποία τελικά καταλήγει να εντοπίσει τις αιτίε των ατυχημάτων. Τα εθνικά δίκτυα λοιπόν υπηρεσιών διερεύνησης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα αποτελεσματικό μέσο το οποίο μας επιτρέπει να καλύψουμε τα διαφορετικά επίπεδα που υπάρχουν όσον αφορά τις υπηρεσίες διερεύνησης σε κάθε κράτος μέλος. Τώρα εδώ θα ήθελα να πάω λίγο πιο μακριά όμως από την πρόταση της Επιτροπής και να ζητήσω να καθοριστεί η αποστολή των δικτύων αυτών και να έχουμε δίκτυα ισχυρά που να μπορούν να δράσουν και να εγγυθούμε την προστιθέμενη αξία που έχουμε από τη δημιουργία τέτοιου δικτύου. Έτσι έχουμε τις τροπολογίες 4 με 6 και 20 με 30 πολλοί φοβούνται ότι τα δίκτυα αυτά αποτελούν ε, ένα βαρύ διοικητικό σώμα. Εδώ όμω θέλω να διευκρινίσω ότι το δίκτυο δεν αποτελεί μια νέα υπηρεσία, ένα νέο οργανισμό, δεν χρειάζεται νέο νομικό καθεστώ, δεν δημιουργούμε δηλαδή ένα επιπλέον διοικητικό όργανο. Εγώ είμαι η πρώτη που δεν θέλω κάτι τέτοιο. Όμω πρόκειται ε, για την βελτίωση δομών που ήδη υπάρχουν, προσφέροντα την αποστολή του, των μονάδων αυτών που ήδη υπάρχουν κάτι παραπάνω. Το δίκτυο λοιπόν δεν αντικαθιστά τα ήδη υπάρχοντα γραφεία διερευνητικά που ήδη έχουμε, αλλά θέλει να τα ενισχύσει και θέλει η κάθε υπηρεσία, η κάθε εθνική υπηρεσία διερεύνησης να μπορέσει πιο αποτελεσματικά να δράσει. Το δεύτερο σημαντικό πράγμα που διακυδεύεται εδώ πολιτικά είναι η στήριξη των θυμάτων και των οικείων τους. Και εδώ παλέρχομαι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που την αναπτύσσω περισσότερο στην έκθεσή μου. Όσον αφορά πρώτα απ' όλα την κατάσταση επιβατών, είναι σημαντικό να υπάρχει προθεσμία, γιατί αλλιώς έχουμε καταχρήσεις και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο για τους πολίτες. Αποφάσισα λοιπόν να διατηρήσω την υποχρέωση Κατάσταση επιβατών εντός τη ώρα που ακολουθεί την αναγγελία ενό ατυχήματο. Και μάλιστα έχω διευρύνει και το επίπεδο εφαρμογής σε αεροπορικές ε, εταιρείε και πτήσεις γενικότερα και όχι μόνο για εκείνες που αναχωρούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για όλες. 10 με 53, 54, 55, 56 αναφέρονται στο θέμα τόμου με το οποίο πρέπει να έρχεται σε επαφή η αεροπορική εταιρεία για να ενημερώσει για το ατύχημα τον οικείο κάποιου θύματος. Πρέπει δηλαδή οι αεροπορικές εταιρείες να προτείνουν στους επιβάτες να δηλώνουν όταν κάνουν την κράτησή τους ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούν να απευθυνθούν ευρωπαϊκές εταιρείε σε περίπτωση ατυχήματο. Εδώ βέβαια τίθεται και το θέμα των προσωπικών δεδομένων. Και γι' αυτό σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο ε, επιθεώρηση Προσωπικών Δεδομένων, ε, συνονιθήκαμε και είπαμε ότι τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τίποτα για εμπορικού λόγου. Επίσης έχω ε, συμπληρώσει και με τις τροπολογίες μου 59 και 60 το σημείο αυτό. Θέλω να δημιουργηθεί μια υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να επαληθεύουν ότι οι αεροπορικές εταιρείες έχουν σχέδιο αντιμετώπισης κρίσης. Εξού και τροπολογία 61 που μιλάει για, την, ε, για τον ορισμό ενός ε, υπεύθυνου για την επαφή με τους οικείους των θυμάτων. Έτσι θα ενημερώνονται οι οικοί των θυμάτων όχι μόνο για το ατύχημα αλλά και για τις διαδικασίες που ακολουθούν. Έπειτα στις τροπολογίες μου 11 και 45 ενισχύω τις διατάξεις που επιτρέπουν στους οικείους των θυμάτων να έχουν πληροφορίες για την ε, διαρευνητική διαδικασία των αιτιών του ατυχήματο και για την ασφάλεια. Τέλος, πάλι για τα θύματα, έχω βάλει εδώ την υποχρέωση όλων των εταιριών που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβουν τη δέσμευση να τηρούν τις διατάξεις της Σύμβασης του Μόντρελ για την αστική ευθύνη του αερομετοφορέα για τις αποζημιώσεις κλπ. Αυτή είναι η τροπολογία μου 62. Ένα άλλο σημείο, το οποίο δεν θίξαμε με κάθε λεπτομέρεια την προηγούμενη φορά και που είναι όμως πολύ σημαντικό, έχει να κάνει με τις ε, εκθέσεις για τα συμβάντα. Εδώ πέρα πρόκειται για ένα κεντρικό αποθετήριο πληροφοριών, το οποίο προορίζεται για να συγκεντρώνει όλα τα περιστατικά που συμβαίνουν εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ δεν χρησιμοποιείται αρκετά. Είναι μια βάση δεδομένων αρκετά ενδιαφέρουσα που αν κάποιος υπεύθυνο οριστεί για την ανάλυση των δεδομένων αυτών, τότε ίσως μπορούμε να αποφεύγουμε τα διάφορα συμβάντα που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά και που κάποια στιγμή μπορεί να οδηγήσουν και σε κάποιο ατύχημα. Μπορούμε λοιπόν να αναρωτηθούμε αν ξέραμε τα προβλήματα αυτά που έχουν προκύψει μέχρι τώρα, ε, ατυχήματα όπως εκείνο του Ρίος που θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Το ίδιο και για το 2005 της εταιρεία Ήλιος. Μήπως και αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχαμε αναλύσει αντίστοιχα συμβάντα στο παρελθόν. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε έτσι να βελτιώσουμε σημαντικά την ασφάλεια των πτήσεων. Τέταρτον, συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας στις έρευνες. Από το 2003 ο οργανισμός αυτός δίνει ε, πιστοποίηση των αεροσκαφών. Είναι λοιπόν λογικό ο οργανισμός αυτός να συμμετέχει και στις διερευνήσεις όσον αφορά την ασφάλεια για να προσφέρει πραγματογνωμοσύνη και πληροφορίες στους διερευνητές. Όμως τα γραφεία, τα διερευνητικά των χωρών μελών που έχουν βέβαια κάποια εμπειρία και συχνά εξαρτώνται από το ίδιο Υπουργείο δεν φτάνουν. Ο οργανισμός θα μπορούσε να προσφέρει κάτι παραπάνω, αλλά δεν έχουν τη συνήθεια να συνεργάζονται μεταξύ τους. Έχει υπάρξει σύγχυση στο παρελθόν για τις διάφορες πλευρές που συμμετέχουν σε μια διερεύνηση ατυχήματος. Το σχέδιο αυτό κανονισμού λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για την συμμετοχή του οργανισμού στις διερευνήσεις ατυχημάτων χωρίς όμως να μπορεί να επηρεάζει ε, την έρευνα ή να εκτελεί εκ άλλη διερεύνηση. Είναι σημαντικό επίσης ο όρος που χρησιμοποιούμε να είναι πολύ συγκεκριμένο στο παράρτημα 13 και νομίζω ότι πάνω σε αυτό όλοι συμφωνούμε και το Συμβούλιο συμφωνεί μαζί μας για το ότι ο οργανισμός που πιστοποιείται αεροσκάφη δεν μπορεί να είναι και κριτής και κρινόμενος. Έχει χρησιμοποιηθεί ο όρος εμπειρογνώμων για τον οργανισμό. Εγώ λέω όμως να αντικατασταθεί ο όρος αυτός από τον όρο σύμβουλος που χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις. Προτείνω λοιπόν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας να έχει δικαιώματα συμβούλου, έτσι όπως καθορίζονται από το παράρτημα 13 της Σύμβασης σχετικά με τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία. Το τελευταίο σημείο μου είναι ο συντονισμός που γίνεται ανάμεσα ε, στην ε, διερεύνηση, την τεχνική και την δικαστική. Εδώ είναι ένα πολύ λεπτό σημείο αυτό και ίσως θα είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο λοιπόν ε, Επιθεώρησης Προσωπικών Δεδομένων, με το οποίο συναντήθηκα και εγώ, πιστεύει ότι η πρόταση κανονισμού δεν πάει αρκετά μακριά όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Και όπως ήδη το είχα πει και στο έγγραφο εργασία μου, εγώ θέλω να προστατεύσω τις ευαίσθητε πληροφορίες και να βρω μια λογική ισορροπία ανάμεσα στην προσωπία των προσωπικών δεδομένων και από την άλλη φορά το δικαίωμα των θυμάτων να έχουν πρόσβαση στι ε, πληροφορίε τη διερεύνηση. Εδώ λοιπόν στην πρότασή μου αυτή νομίζω ότι ευθυγραμμίζομαι καλύτερα με την γνωμοδότηση του Γραφείου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και λέω ότι όλα όσα ε, δίνονται στα θύματα και τους οικείους τους να έχουν να κάνουν με γεγονότα βάσει της παραγράφου 15 α, β και γ και να δίνονται προς την ε, δικαιοσύνη μόνο ε, συγκεκριμένα στοιχεία όπως λέει η τροπολογία μου 40, ό,τι αφορά δηλαδή τη διαπίστωση των γεγονότων και την ανάλυση των τεκμηρίων να πρέπει να διαβάσετε στη δικαιοσύνη, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία θα πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά. Εν κατακλείδη. Έχω συντάξει και ένα ειδικό άρθρο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είναι τροπολογίες 12, 56 δεύτερο τμήμα και 63 με 65. Αυτές λοιπόν, όσο πιο γρήγορα μπορούσα, σας έδωσα τις κατευθυντήριες γραμμές. Ελπίζω ότι και εσείς με τις δικές σας προτάσεις θα βελτιώσετε ακόμα περισσότερο το κείμενό μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Ντεβεράκ. Τώρα, η Σκιώδης. Από τους σοσιαλιστές πρώτα, ο κύριος Ζένκιν. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποια σχόλια που έχουν ως εξής. Η ομάδα μας θα στηρίξει τον κανονισμό αυτόν. Πιστεύουμε ότι είναι ένα σημαντικός κανονισμός και αναγκαίος κανονισμός. Οι τροπολογίες της εισηγήτριας πιστεύουμε ότι πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και απορρέουν εξάλλου και από τις συζητήσει και τους συμβιβασμού στους οποίους καταλήξαμε μέχρι τώρα. Γενικά μιλώντας λοιπόν συμφωνούμε. Τώρα, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Εμείς στην Πολωνία έχουμε τις δικές μας εμπειρίες. Διερευνούμε το μεγάλο αεροπορικό ατύχημα που έλαβε χώρα στην πολιτική αεροπορία. Γίνεται ανάλυση, συζητάμε το θέμα και πιστεύω ότι εδώ μπορούμε να καταλήξουμε σε μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Και θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποια πρακτικά ζητήματα. Συμφωνώ απόλυτα για το ότι ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να διασφαλίζει την ανεξαρτησία της διερεύνησης των ατυχημάτων. Όταν όμως γίνεται ένα ατύχημα, η σχετική αρμόδια επιτροπή αρχίζει να δουλεύει. Συγχρόνως όμως το γραφείο της εισαγγελία από τη δικιά του την πλευρά προχωράει επίσης σε μια έρευνα. Οπότε βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει σύγκρουση εξουσιών. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την εισηγήτρια μάλλον να ζητήσω από την εισηγήτρια να συμπεριλάβει κάτι τονίζοντας την ανεξαρτησία του διαρευνητικού οργάνου και το γεγονός ότι η εισαγγελία κάνει τη δικιά της έρευνα δεν πρέπει να επηρεάζεται η διερεύνηση του ατυχήματος η οποία βρίσκεται να εξελίξει. Διότι αλλιώς μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου ορισμένοι ερευνητές να μην δίνουν πληροφορίες. Μετά την διερεύνηση πάντως του ατυχήματος, όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται να μεταφερθούν να πηγαίνουν στις αρμόδιες αρχές. Και όλα τα προσωπικά δεδομένα να προστατεύονται. Τα δεδομένα δηλαδή εκείνα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την έρευνα αυτή καθεαυτή του ατυχήματος. Ε, κατά τα στηρίζω την ε, πρόταση της εισηγητρίας. Ε, ο κύριος Κατσίνα από την Άλντε τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει και για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με, την, με το πρώτο σχέδιο λαμβανωμένων υπόψη των ε, πρόσφατων τροπολογιών οι οποίες ε, βοηθούν ε, μας βοηθούν στην κατανόηση και στην εμάθηση της συστηματικής προσέγγισης αυτού του ζητήματος. Εγώ θεωρώ πως στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα είμαστε σε θέση να θεσπίσουμε μια νέα νομοθεσία η οποία θα βοηθήσει πολύ την ασφάλεια των αερομεταφορών. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω είναι η λίστα των τροπολογιών η οποία μας υποβλήθηκε από την European Cockpit Association ε, όπως ε, και από τις ε, Διεθνείς Ενώσεις των Ελεγκτών Εναερίας Κυκλοφορίας που ζητούν να αναφέρονται σε εθελοντική βάση τα διάφορα συμβάντα ε, και να ζητούν εξηγήσει σε ό,τι αφορά ατυχήματα τόσο οι πιλότοι από τη μία πλευρά όσο και ελεκτές ενέργειες κυκλοφορίας από την άλλη να ζητούν περισσότερες οδηγίες ε, και ούτω καθεξής. Θα ήθελα να ρωτήσω την εισηγήτρια ποια είναι η δική της γνώμη σε σχέση με αυτές τις προτινόμενες τροπολογίες, οι οποίες είναι πολύ συστηματικές και κατευθύνονται προς τον καλύτερο έλεγχο από την πλευρά των ελεκτών και κυκλοφορίας, ούτως ώστε να θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο, να μην θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο εκ των προτέρων ένοχοι από τους η ε, ε, γενικά από το δικαστικό σύστημα. Θα ήθελα να ξέρω από την εισαγγελία ποια είναι η δική τη ε, θέση και τη θεωρία εκείνη πώς θα πρέπει να γίνει στο μέλλον. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε για του πράσινου η κυρία Νίχτεμπεργκ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Το βασικό πρόβλημα το οποίο εντοπίζεται σε σχέση με αυτή την έκθεση και η έκθεση κάνει κάποια βήματα για την επίλυση αυτού του προβλήματος είναι να μην υπάρξουν κολλήματα σε ό,τι αφορά την κανονική ε, δίκαστη ε, διαδικασία, αλλά από την άλλη πλευρά να είμαστε σε θέση να βρίσκουμε σημεία τα οποία είναι, ε, παρουσιάζουν λάθη μέσα σε, στις σχετικές διαδικασίες και το να επιτύχουμε την ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο στοιχεία είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή από τη μία να μην έχουμε παρακόλληση της δικαιοσύνης και των διάφορων ερευνών και από την ε, άλλη ε, πλευρά να μην έχουμε την εξαίρεση από, όλη την, ε, από όλες τις σχετικές έρευνες συγκεκριμένων λεπτομεριών οι οποίες είναι σημαντικές. Για μένα το κυρίω ζητούμενο εδώ είναι να είμαστε θέσει να προστατεύσουμε τους δυνητικούς whistleblowers, δηλαδή εκείνους οι οποίοι θα κοινοποιήσουν τέτοιου είδους παρατυπίες. Δηλαδή, εάν κάποιοι επιθυμούν να αναφέρουν κάποια στοιχεία τα οποία από συστηματική άποψη είναι πολύ σημαντικά χωρίς να σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο συμβάν, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα απολέσουμε πολύ σημαντικές ε, πηγές πληροφόρησης. Άρα λοιπόν η προστασία αυτών των ατόμων, των whistleblowers, είναι πολύ σημαντική μέσα στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι η προστασία των δεδομένων. Και εδώ πάλι τίθεται ένα ζήτημα ισορροπίας. Να θυμίσω ότι μετά από το τσουνάμι για παράδειγμα, στην Νοτιοανατολική Ασία, είχε προκύψει για πολλές οικογένειες ε, το πρόβλημα ότι μετά από πιέσεις που ασκήθηκαν από διαφόρους δεν αναφέρθηκαν τα ονόματα των οποίων είχαν επιστρέψει γιατί θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται γιατί εκεί πάρα πολύ η, σχετικά μεγάλος αριθμός τουριστών. Άρα λοιπόν υπάρχουν συμβατά τα οποία συμβαίνουν μέσα σε κάποιες γενικότερες προϋποθέσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε εκτεταμένες ε, συζητήσεις δημόσιες. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε προστασία των δεδομένων των ε, ατόμων που εμπλέκονται σε τρία συμβάτα και ε, να διασφαλίσουμε την προστασία των οικογενειών. Από την άλλη πλευρά, το να έχουμε ένα πρόσωπο για επαφές εκ των προτέρων Ε, σε ό,τι αφορά τα ίδια τα δεδομένα κράτησης ε, ε, ήδη είναι κάτι το προβληματικό γιατί αυτό τροφοδοτείται μέσα στο ΣΥΡΙΣ και κατά συνέπεια οι Αμερικανικές αρχές έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Είναι σαφές κάτι τέτοιο και κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στη δική μου αντίληψη σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Άρα λοιπόν για μένα θα είναι πολύ δύσκολο να βρούμε μια λύση. Από τη μία πλευρά δηλαδή να αναφέρουμε ένα τέτοιο πρόσωπο, από την άλλη όμως ε, πλευρά κάτι τέτοιο να ε, περιλαμβάνεται μέσα στα δεδομένα τα οποία μετά μεταβιβάζονται στις ε, αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών ως πακέτα. Κάτι τέτοιο δεν μας αρέσει γιατί ενδεχομένως εκεί θα μπορούν να περιλαμβάνονται και ευαίσθητου χαρακτήρα πληροφορίες. Θα πρέπει να τις προστατεύσουμε λοιπόν. Και ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς το τι ακριβώς θα κάνουμε σε αυτό το τομέα. Θεωρώ πως ε, θα πρέπει να επανεξετάσουμε αυτό το ζήτημα του μη διαχωρισμού των σχετικών ε, δεδομένων κράτησης όπως καταγράφονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς προφανώς θα συζητήσουμε εκ των προτέρων τις τροπολογίες μας με την εισηγήτρια γιατί ε, συνολικά έχει θέση με πολύ σωστό ε, τρόπο το όλο ε, πρόβλημα και θεωρούμε πως μπορούμε να βελτιώσουμε λίγο ακόμα την εκθέση. Ευχαριστούμε την κυρία Τίθεμπεργκερ, γνώση της Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κυρία γιατί προσπάθησε να μας συγκεντρώσει για να συζητήσουμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, αλλά δεν τα καταφέραμε τελικά να συζητήσουμε. Ε, λοιπόν, δεν θα διατρέξω όλες τις τροπολογίε, αλλά όπως ήδη αναφέρθηκε, καλύπτει ε, μια σειρά από σημεία ε, τα οποία θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω. Ε, θα πρέπει να εξετάσουμε το κατά πόσο είναι καλές οι δικές μας έρευνες ε, σε ό,τι αφορά τα αντιχήματα. Ναι, ήταν ε, καλής ποιότητας μέσα στις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, αλλά η επιτυχία του βασίζεται του ότι ήταν ανεξάρτητες αυτές οι έρευνες και κρατάω και το σχόλιο του Πολωνού συναδέλφου ότι δηλαδή θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι ανεξάρτητες αυτές οι έρευνες και μένουν και ανεξάρτητες από την από τον ε, τομέα της δικαιοσύνης από την ε, δικαστική τομέα. Ελπίζω λοιπόν να μην χρειαστεί να κάνουμε κάτι για να αποτρέψουμε ε, κάτι τέτοιο. Τώρα, σε ό,τι αφότερα σχόλια, η κυρία Τιβεράκ, νομίζω πως έχει δίκιο όταν θίγει το ζήτημα των θυμάτων. Λέμε ότι οι σχετικέ πληροφορίε στα δεδομένα θα πρέπει να διαβάζονται μέσα σε μία ώρα. σω η μία ώρα να μην είναι κάτι το ρεαλιστικό. σω θα πρέπει να λέμε το ταχύτερο δυνατό να είμαστε πιο πραγματιστέ, γιατί με την τεχνολογία πάντοτε είναι δυνατόν να υπάρξει περισσότερη πρόοδο, να υπάρχει ταχύτερη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών. Ε, τώρα, ε, συμφωνώ με την κυρία Λίχτεμπεργκερ και με το πρόσωπο επαφή και την αναφορά αυτού του προσώπου στα δεδομένα κράτηση. Συμφωνώ ε, μαζί τη. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πρακτικό κάτι τέτοιο, βέβαια, λύση προτείνεται από την πλευρά τη, αλλά ίσω θα πρέπει να το συζητήσουμε με του εμπλεκόμενου τώρα σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα της, ε, των προτέρων ενοχή, ας το πούμε έτσι, δηλαδή το πώ ε, απευθύνονται κατηγορίε ε, στου πιλότους, στο πλήρωμα και ούτω καθεξή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ χρήσιμο. Αυτό προέκυψε μέσα από τις συζητήσεις στο ΘΥΙ και η συγγήτρια. Ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε εξεχωριστά στο πλαίσιο δηλαδή άλλου κανονισμού σε ό,τι αφορά την υποβολή εκθέσεων, σε ό,τι αφορά την, ε, την ε, τέτοιου είδους συμβάτα, δηλαδή τον, την συχνότητα τέτοιων συμβάτων. Και ενδεχομένω θα πρέπει εκεί να ε, περιλάβουμε και την εθελούσια αναφορά, την εθελούσια ενημέρωση, γιατί εκεί θίγεται και όλο το ζήτημα αυτό των whistleblowers, δηλαδή των ατόμων που επιθυμούν εθελούσια να ενημερώσουν. Ε, δεν είναι ακριβώς ε, whistleblowers, δηλαδή ε, είναι απλά κάποια άτομα τα οποία έχουν τη βούληση να, φέρουν ότι μέσα στην γραμμή των εντολών, μέσα στην γενικότερη διοίκηση υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν λειτουργούν σωστά. ένα τελευταίο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω αφορά την Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτό το σχέδιο και έγιναν πάρα πολλέ προσπάθειες και πολλή δουλειά για να βελτιωθεί. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα σχόλια που κάνουμε. Ε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένοι ε, ευθύ εξ αρχή με τον τρόπο που η έκθεση εκείνη συντάχθηκε ευθύ εξ αρχή. Εκπονήθηκε δηλαδή με έναν τρόπο ε, που δείχνει ότι κάποιος δεν ε, εξέτασε από κοντά το πώς γίνεται μια τέτοια έρευνα. Ε, μιλάμε για ένα τεχνικό κανονισμό και κατά συνέπεια η διάρθρωσή του θα πρέπει να ε, συνάδει και λίγο με ε, το αντίστοιχε νομοθεσίε και αλλού και σε διεθνέ επίπεδο υπάρχει συνεργασία και με τρίτες χώρες και νομίζω πως η αντίστοιχη ομάδα εργασία του Συμβουλίου έχει ξεκινήσει κάποιε εργασίε παράλληλα με εμά. και έχω ρίξει μια ματιά στο σχετικό κείμενο του Συμβουλίου, έχει αλλάξει την ε, σειρά των διαφορετικών ε, άρθρων, ε, περιλαμβάνει μία σειρά από αλλαγές, είναι καλύτερα εκπονημένο και παρότι προφανώς θα μπορούσε να βοηθηθεί περισσότερο με τις τροπολογίες όπως αυτές της κυρίας Ντεβεράκη, είναι πολύ καλύτερο από το αρχικό σχέδιο. και προφανώ βέβαια αυτό το κείμενο θα πάει και με τι ε, δικέ μα τροπολογίε και τι τροπολογίε ε, τη κυρία Σάντεβερακ στο Συμβούλιο. Για να προσπαθήσουμε τελικά να επιτύχουμε μια συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση, σα λέω όλη η διάρθρωση, όλη η δομή αυτού του κειμένου αυτή τη ε, έκθεση θα πρέπει να τροποποιηθεί. Ε, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ πω συνολικά θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια καλή συμφωνία αλλά θα ήθελα να ακούσω κάποιο σχόλιο από την πλευρά τη Επιτροπή όταν πάρει το λόγο. Ω προ αυτέ τι παράλληλε εργασίε που συμβαίνουν, δηλαδή από τη μία πλευρά εδώ και από την άλλη πλευρά στο Συμβούλιο. Ε, Ο κύριο Γκρό, ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω εγώ καταρχήν την εισηγήτρια για τι ε, εργασίε τη ε, πράγματι διάφορες παρατηρήσει δείχνουν ότι έχουμε εδώ να κάνουμε με έναν ευαίσθητο τομέα και από την άλλη πλευρά διαπιστώνουμε ότι η διάρθρωση εδώ αυτού του τομέα αδιαφέρει ανά ε, ο κράτος μέλος ε, κατά συνέπεια είναι δύσκολο να βρούμε μια κοινή ετοδομή. Ε, τα τρία βασικά στοιχεία κατά τη δική μου άποψη, τρεις βασικές προϋποθέσεις είναι πανευρωπαϊκός χαρακτήρας, ανεξάρτητες και ε, ανάληψη, δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας. Ε, δηλαδή ε, δεν θα πρέπει μόνο να διαπιστώνεται το γιατί συνέβη ένα ατύχημα αλλά να υπάρχει δυνατότητα αυτό ο μηχανισμός να δίνει κάποιες συστάσεις εκ των προτέρων για την αποφυγή δηλαδή ατυχημάτων. ούτω ώστε να μην έχουμε δηλαδή εκ των προτέρων διαβίβαση τέτοιων ε, πληροφοριών, οι οποίε ε, ήδη από τώρα υπάρχουν κάποια στοιχεία για αυτέ, ε, υπάρχουν κάποιε ενδείξει για αυτέ τι πληροφορίε. εάν δεν έχουμε μια τέτοια προσέγγιση θα έχουμε την, τον κίνδυνο και να υπάρχει διαφορετική δομή ένα κράτος μέλος και από την άλλη πλευρά εκείνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν κάποιες να δώσουν κάποιε ε, πληροφορίε δεν θα ήταν σε θέση να το κάνουν ή θα απέφευγαν να το κάνουν γιατί θα φοβούνται ότι ενδεχομένω θα εμπλακούν σε μια δικαστική διαδικασία, θα βρεθούν κατηγορούμενοι και ούτω καθεξή. Ε, και εδώ προσπαθούμε ουσιαστικά να ε, προσανατολιστούμε με με ένα παρόμοιο τρόπο στα όσα συμβαίνουν στον τομέα των συνδρομικών μεταφορών ε, και δεν είναι θετικό αυτό γιατί εδώ θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη ανεξαρτησία σε ό,τι αφορά τις έρευνες. Ε, η ε, συγκίτρια έχει καταφέρει να επιτύχει εδώ μια ισορροπία ανάμεσα αφενός στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και από την άλλη την ανθρώπινη, πούμε, διάσταση. και θεωρώ και εγώ πως με αυτήν την νέα πρόταση θα κάνουμε ένα βήμα μπροστά ε, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τα οποία ε, θίγουμε με αυτές τις τροπολογίες συγκεντρώνουν την ε, σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας εδώ σε αυτή την αίθουσα ως προς το πώς φανταζόμαστε τα πράγματα, το πώς θέλουμε να κινηθούν αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι συμφωνεί το Συμβούλιο μαζί μας και από εκεί και μετά ε, είμαστε αρκετά θαραλέοι για να κάνουμε αυτό που είδαμε να συμβαίνει μεταξύ άλλων στη Ουάσιγκτον όπου δηλαδή η σχετική έρευνα ήταν πραγματικά ανεξάρτητη, ακόμα και από, πολιτικό, ε, ε, από πολιτικής πλευράς ανεξάρτητη, και ότι είχε τους κατάλληλους πόρους και μάλιστα κανένας δεν είχε το θάρρος να, να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα τέτοιων ερευνών, γιατί ε, πραγματικά ήταν ανεξάρτητες. Εάν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, πραγματικά θα έχουμε κάτι, καταφέρει κάτι το πολύ χρήσιμο και για τους πολίτες μας. Δύο παρατηρήσεις θα κάνω κι εγώ. Ε, πέρα από τα συγχαρητήρια. Τα πεθαίνω κι εγώ. Ε, για αυτές τις προτάσεις. Τώρα σε ό,τι αφορά την τοπολογία δοθώ και μετά σε ό,τι αφορά την διαγραφή του άρθρου 15 παράγραφος 3 για την επανεσαγωγή του άρθρου 21 γίνεται μια προσπάθεια να υπάρχουν, να, να βάλουν χώρα με καλύτερο τρόπο διάφορες έρευνες ε, στην Ευρώπη και αυτό θα βοηθήσει βέβαια και στην αποτροπή αντίστοιχων ατυχημάτων λόγω ε, προβλημάτων σε ό,τι αφορά τα υλικά. Ε, σε αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιμείνουμε. Το δεύτερο που θα ήθελα να θίξω ε, αφορά την ΕΑΣΑ και πρόκειται και για ερώτηση. Σε σχέση με τη συζήτηση που έγινε και χθες σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς, να πω ότι εδώ έχουμε ένα παράδειγμα. Εάν ρίξουμε μια ματιά στην πραγματικότητα σήμερα, αξίζει τον κόπο να εξετάσουμε το καθώς σε ό,τι αφορά τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και έχει νόημα να συζητήσουμε τέτοιου οργανισμού για τα κράτη-μέλη. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι η ΆΣΑ δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να επηρεάζει με κανένα τρόπο τι έρευνε, οι οποίε θα χώρα. Θα πρέπει να είναι σαφέ στην Επιτροπή μα. ότι η ΆΖΑ θα πρέπει να συμμετέχει με καθεστώ παρατηρητή σε τέτοιου είδου έρευνε. Και δεν θα πρέπει να παρεκκλίνουμε από αυτό στο πλαίσιο των περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, τίθεται σε αυτό το πλαίσιο ένα ερώτημα. Καθώς ε, η ΆΖΑ έχει αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες εδώ πρωτοβουλίας, θα πρέπει να συμμετέχει ως ε, πιστοποιημένος ε, εκπρόσωπος σε μια σχετική έρευνα, τουλάχιστον σύμφωνα με την Σύμβαση του Σικάγο. Αλλά στο άρθρο 10 της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι οι εθνικές αρχές ερευνών είναι εκείνε οι οποίε ορίζουν τον εκπρόσωπο σε ό,τι αφορά δηλαδή, την αρμοδιότητα και την ανάληψη πρωτοβουλία. Άρα δηλαδή θα πρέπει να ορίζεται από τη δική του πλευρά ένα εκπρόσωπο τη. ΕΑΣΑ. Οπότε θα ήθελα να ξέρω, ε, δεν ξέρω ή από εσάς ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να λάβω μια απάντηση, αν ερμηνεύω σωστά αυτό το σημείο, ε, αυτό το άρθρο 10, δηλαδή ή αν λύνεται με κάποιο άλλο τρόπο αυτό το πρόβλημα. Η απο εσα η απο την ευρωπαικη επιτροπη θα ηθελα να λαβω μια απαντηση αν ερμηνευω σωστα αυτο το σημειο αυτο το αρθρο 10 δηλαδη η έχει το, το λόγο. Ε, κύριε Τιβεράκ, ε, πραγματικά όλοι το είπαν, θα το πω και εγώ, βελτιώσατε πολύ, κατά πολύ αυτή την πρόταση την οποία λάβαμε. Ακολουθείτε τη σωστή κατεύθυνση. Δύο σύντομα σχόλια θα κάνω σε ό,τι αφορά ε, τα προσωπικά δεδομένα. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Λίχτεμπεργκερ, δηλαδή θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε σχέση με το τι συμβαίνει με την μεταβίβαση των δεδομένων από ε, πτήσει, ε, πράγμα το οποίο συζητείται αυτή την περίοδο και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Εκείνο που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι ο στόχο. Ποιο είναι ο στόχο αυτή τη έκθεση που συντάσσεται είναι να διαπιστώνεται ακριβώ η αιτία των αεροδρομικών ατυχημάτων. Άρα λοιπόν δεν συμφωνώ σε αυτό το σημείο με την κυρία Γκρόση. Θα πρέπει να γνωρίζουμε, ναι, έχει νόημα να γνωρίζουμε γιατί συνέβη κάτι τέτοιο. Μόνο αν το γνωρίζουμε θα μπορούμε στο μέλλον να αντλούμε κάποια συμπεράσματα και να ε, προβαίνουμε σε μια πρόληψη. Θέλουμε λοιπόν να διαπιστώνουμε τις αιτίε και να προστατεύουμε τους επιβάτες και προφανώς όλο το επίπεδο από μελλοντικά ατυχήματα. Για να διαπιστώνουμε τις αιτίε χρειαζόμαστε αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως. Δηλαδή πρώτον ανεξαρτησία της αρχής που είναι αρμόδια για την έρευνα. Το είδαμε στην ε, Ουάσιγκτον πόσο ε, πόσο μεγάλη είναι η ανεξαρτησία αναφέρθηκε ήδη ότι υπάρχει και, και από πολιτική άποψη ανεξαρτησία και σε αυτό συγκαταλέγεται ε, το να αποφεύγεται η διαβίβαση ε, πληροφοριών στο ευρύ κοινό από νωρίς. Δηλαδή ε, κάποιε αρκετέ πληροφορίε οι οποίε δίνονται ότι ενδεχομένω δηλαδή να επρόκειτο για από την πλευρά του πιλότου ή για ένα μήνο ε, που λιώνει οτιδήποτε άλλο. Μπορεί κάτι τέτοιο να ισχύει, αλλά τελικά ε, ενδέχεται και να μην ισχύει. Ταυτόχρονα, πραγματικά υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν, το, για παράδειγμα και εγώ αν ήμουν πιλότος δεν θα ήθελα να πω Ακριβώ ε, πω κάτι θεωρουσα πω κατι τετοιο θα μπορούσε να με ε, θέσει στην ε, θέση του κατηγορούμενου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ συγχαίρω την κυρία Ντεβιράκ, όπως πάντα συμβαίνει με τις εκθέσεις της, έτσι και τώρα, είναι λιτές και σοβαρές. έχω δύο πράγματα που με απασχολούν και η συγγήτρια τα χειρίζεται καλά. Τα έχει εντοπίσει και η ίδια και έχει εκφράσει τις ανησυχίες της. Το ένα είναι η προστασία προσωπικών δεδομένων. Και θέλω να επιμείνω πάνω σε αυτό. Γιατί υπάρχει κάπως σύγκρουση ανάμεσα στις πληροφορίες της διερεύνησης της πολιτικής αεροπορίας με τις ε, νομικές έρευνες. Προσοχή λοιπόν, κάτω από τι όρους γίνονται και ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των πρώτων, μπορεί να οδηγήσουν σε προσφυγές που δεν είναι επιθυμητές. Δεύτερον, πρέπει να προσπαθήσουμε, και το κάνει και η κυρία Βεράκ, αλλά Έχω υπάρξει δικηγόρο σε περιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων και ξέρω ότι γίνονται πάρα πολλέ προσφυγέ ε, για τέτοια θέματα. Δεύτερον, η στήριξη των θυμάτων. Εποφελούμαστε από τα μεγάλα ατυχήματα που είχαμε στην Ευρώπη αρκετά πρόσφατα για να αναλύσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη στήριξή μας στα θύματα. Πρέπει να διευκολύνουμε όσον αφορά τα θύματα και βέβαια μιλάω και για τους οικείους των ε, θυμάτων που έχουν ε, χάσει τη ζωή τους. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να τους ενημερώνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα για τον κατάλογο των επιβατών. Και εδώ γίνονται προσφυγές συχνά επειδή καθυστερεί η διαδικασία ε, μέσω του DNA των ε, θυμάτων για να ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Δηλαδή πρώτα έχουμε τον κατάλογο των επιβατών και μετά βέβαια έχουμε την έρευνα του DNA για να εντοπίσουμε ακριβώς ε, τα θύματα στο χώρο του ατυχήματος. Για άλλη μια φορά συγχαίρω την εισηγήτρια. Έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και ελπίζω σύντομα να έχει ολοκληρωθεί αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ. Η κυρία Άλβαρης έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την κυρία Ντεβιράκ. Την ευχαριστώ για την έκθεσή της. Υπάρχουν εδώ πολλά ζητήματα που έχουν ε, τεθεί και την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα μόνο. Στην πρόταση της Επιτροπής και που η κυρία Ντεβιράκ στην έκθεσή της ε, περιλαμβάνει ως τροπολογία για να οριστούν καλύτερα ή να οριστεί καλύτερα η αποστολή του οργανισμού, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας. Εγώ λοιπόν θα έλεγα ότι πρέπει να πάει ακόμα πιο μακριά στην αποστολή αυτή και να βάλει και την ευθύνη πιστοποίησης γιατί έτσι πιστεύω ότι βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η διαρευνητική αποστολή. Επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν ε, επικαλύψεις. Ό,τι κάνουν οι εθνικές αρχές δηλαδή, να μην υπάρχει επικάλυψη και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. στο δίκτυο πρέπει να υπάρχει και υποχρέωση στήριξης των θυμάτων και των οικείων τους. Έρχομαι τώρα στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας. Εδώ συμφωνώ με όσα υπόθηκαν ήδη, ότι δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι και κριτής και κρινόμενος. Πρέπει να εγγυθούμε εδώ για την διερευνητική διαδικασία ότι θα είναι ανεξάρτητη. Στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώνω ότι δεν είναι ξεκάθαρο. Μιλάμε εδώ για τα δικαιώματα του οργανισμού και όχι για τις υποχρεώσεις του οργανισμού. Ένα άλλο στοιχείο κλειδί που δημιουργεί πρόβλημα από ό,τι καταλάβαμε μέχρι τώρα είναι η πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία και η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κακώς έχει την ίδια μεταχείριση όσον αφορά την χρήση των ε, δεδομένων και την δημοσιοποίησή τους. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση. Άλλο, η δημοσιοποίηση για την οποία πρέπει να προβλέψουμε πολύ περιοριστική χρήση μόνο όταν είναι εντελώς αναγκαίο και άλλο είναι η πρόσβαση στα δεδομένα των ερευνητών που πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση για να κάνουν τη δουλειά τους. και να μπορούν να εμβαθύνουν στην διερεύνηση του ατυχήματος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει διάκριση όταν μιλάμε για την στήριξη και άλλο είναι η περίπτωση διαχείρισης κρίσης. Άλλη είναι η δουλειά δηλαδή, που κάνει η αεροπορική εταιρεία σε αυτή την περίπτωση και άλλη είναι ο άλλος είναι ο χειρισμός που κάνουν τα κράτη μέσω μιας διαχείρισης κρίσης. Ήμουνα παρούσα το 2006 όταν ε, οι οικοί περίμεναν τη Ισπανέα την πτήση. Και έτσι από πρώτο χέρι ξέρω την αγωνία τους περιμένοντας τον ε, κατάλογο επιβατών. Πρέπει αμέσως μόλις έχει συμβεί ένα ατύχημα οι αρμόδιες αρχές να έχουν τον κατάλογο επιβατών. γιατί έτσι μειώνουμε κάπως την αγωνία των ανθρώπων που περιμένουν τους δικούς τους. Αλλιώς υπάρχει ανασφάλεια. Θα υποβάλω λοιπόν μια τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση. Και για αυτό που λέγατε για να υπάρχει ένα πρόσωπο επαφής και αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό και θετικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ. Πολλές από τις τεχνικές πλευρές έχουν ήδη σχολιαστεί εδώ. Πρέπει να ενισχύσουμε το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν γίνεται μια ανεξάρτητη διερεύνηση και διάφανη, ενισχύεται η αξιοπιστία της διερεύνησης. Και για τον υπάρχει άτομο επαφής, συμφωνώ ότι πρέπει να ορίζουμε κάθε φορά που παίρνουμε το αεροπλάνο ε, Ποιο θα πρέπει να ειδοποιηθεί σε περίπτωση ατυχήματος. Έχουμε δει να γίνονται ατυχήματα και διαπιστώνουμε ότι οι οικοί υποφέρουν πάρα πολύ, ξέροντας ότι εμπλέκεται στο ατύχημα κάποιος δικός τους. Γι' αυτό ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να υποφέρουν λιγότερο οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να το κάνουμε. Να συμπεριλάβουμε λοιπόν τη διάταξη αυτή ότι πρέπει να υπάρχει, έχει καθοριστεί ένα άτομο, αλλά να υπάρχουν και κάποια πρωτόκολλα επικοινωνίας. Να μην μαθαίνουμε δηλαδή από τα μέσα ενημέρωσης ότι έχει γίνει ένα τύχημα και κάποιος δικός μας έχει χάσει τη ζωή του. Όχι, να υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ξέρω ότι είναι περίπλοκο, αλλά πρέπει να προβληματιστεί η Επιτροπή μας γι' αυτό. Μήπως μπορούμε να καθορίσουμε λοιπόν έναν κώδικα διοντολογίας με τα μέσα ενημέρωσης των κρατών μελών, ώστε όταν γίνεται ένα τύχημα να χειρίζονται την υπόθεση σωστά. Αν δούμε πώς μεταφέρονται τα νέα αυτά στη μία και στην άλλη χώρα, οι διαφορές είναι τεράστιες. Πράγμα το οποίο οδηγεί στο να υποφέρουν ε, τα θύματα και δικοί τους τρεις και τέσσερις φορές παραπάνω. Να το σκεφτούμε λοιπόν. Η νομική αρχή από την άλλη μεριά, εφόσον χρειάζεται, πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία τα οποία της χρειάζονται. Και γιατί, γιατί έχουμε περιπτώσεις κοντά μας που επειδή δεν έγινε αυτό, καταλήγουμε στο να μην καταλαβαίνουμε τις αποφάσεις που λαμβάνονται, να λαμβάνονται στο σκοτάδι, πράγμα το οποίο, το οποίο δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα στις οικογένειες, οι οποίες πρέπει μετά να κάνουν προσφυγές για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που θέλουν. Και έτσι για χρόνια ξοδεύεται χρήμα, γίνονται προσφυγές, χάνεται ενέργεια και προκαλούν πολύ πόνο τέτοιες λανθασμένες διαδικασίες. Πρέπει λοιπόν στο ευρωπαϊκό επίπεδο να συμπεριλάβουμε και μια τέτοια ρύθμιση. Ευχαριστώ πολύ. Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να, να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεση. Είναι πολύ καλή και ας μιλήσουμε. Μιλάμε για ατυχήματα και τα συζητούμε αφού συμβούν. Πολύ συχνά τα ατυχήματα συμβαίνουν και έχουμε και κάποια σχεδόν ατυχήματα, δηλαδή όταν σχεδόν συγκρούνται δύο αεροπλάνα και αποφεύγεται η σύγκρουση τελευταία στιγμή και πρέπει να ερευνούνται αυτά τα επεισόδια. Αν υπάρχουν προβλήματα κατά την πτήση, αν υπάρχουν επί του εδάφους προβλήματα, αν υπάρχουν συστημικά προβλήματα που οδηγούν στα ατυχήματα. Η ΕΑΣΑ λοιπόν θα πρέπει να μαζεύει στατιστικά στοιχεία Όσον αφορά αυτά τα σχεδόν ατυχήματα, όταν μόλις την γλιτώνουν τα αεροπλάνα το ατύχημα. Θα πρέπει να έχουμε και γκρίζους καταλόγους. Αεροπορικών εταιριών, αεροδρομίων, που εμπλέκονται σε αυτά τα επεισόδια, αυτά τα ιωνία ατυχήματα. Να πω και εγώ μερικά λόγια πριν παρεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. αντιδρώ σε αυτά που είπε η κυρία Μπιλμπάου για δεντολογικό κώδικα όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης. Καλή τύχη στη θαυροφορία σας, αυτό έχω να σας πω. Νομίζω ότι είναι καταδικασμένη η προσπάθεια σε αποτυχία. Ποιο πρόβλημα έχουμε στον τομέα των 24 ώρων δελτίων ειδήσεων. Όλοι θέλουν να είναι οι πρώτοι. Τα ειδησογραφικά πρακτορία θέλουν να είναι οι πρώτοι να πούν κάτι και να το ανακοινώσουν. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι αν δεν τους δώσουμε πληροφορίες, ε, εφευρίσκουν πληροφορίες, διότι πρέπει να τροφοδοτούν τις ειδήσει. Το ίδιο ισχύει και με τις εφημερίδες. Θέλουν να πουλούν εφημερίδες, φύλλα και όχι να παρουσιάζουν τα πραγματικά γεγονότα που αφορούν ένα συγκεκριμένο ατύχημα. Και το πρόβλημα είναι να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία. Πόσες πληροφορίες πραγματικά χορηγείς που σταματούν τον εφευρίσκονται πληροφορίες, αλλά πώς πληροφορίες δίδουν, δίδεις και προσέχεις να αντιμετωπίσεις σωστά τα θύματα. Και δεν μιλώ μόνο για επιβάτες. Να τις σωστές πληροφορίες και να μην μαζεύουν, να μην παίρνουν πληροφορίες από τις ειδήσει. Μου αρέσει η προσπάθειά σας, καλός οδοντολογικός κώδικας, καλή τύχη. Θαύματα χρειάζονται κάποιο χρόνο, περισσότερο χρόνο, τέλος πάντων, καλή τύχη. Και κάτι άλλο που θα έπρεπε να πούμε. Η κυρία Ντεβεράκ έχει κάνει μια έξοχη έκθεση. Ξεκινώ από εκεί. Οι αεροπορικές μεταφορές είναι πολύ ασφαλείς. Εύκολα μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για διάφορα μονομένα ατυχήματα πριν γνωρίζουμε που βρισκόμαστε και όλοι πιστεύουν ότι πέφτουν από τον ουρανό συνέχεια τα αεροπλάνα και δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι αεροπορικές μεταφορές είναι ασφαλέστερος τρόπος μεταφοράς. Εμείς θέλουμε να παραμείνει έτσι η κατάσταση. Όμως υπάρχουν θέματα που σχετίζονται με τα μέσα ενημέρωση που ανέφερα. Πρέπει να αποφευχθεί η ιδιαίτερη αυτή αρχή που υιοθετούν τα μέσα ενημέρωση. Ότι αν αμφιβάλλεις για κάτι κατηγόρησε τον πιλότο ή κατηγόρησε τον οδηγό, τον μηχανοδηγό αν είναι τρένο. Διότι θέλουν κάποιο θύμα, ε, κάποιον να κατηγορήσουν. Είναι η κουλτούρα του κατηγορώ αν θέλετε, του κατηγορητηρίου. Αλλά εγώ πιστεύω ότι κάποιο είναι αθώο μέχρι αποδείξει του αντιθέτου και αυτή η αρχή θα πρέπει να εφαρμόζεται, πάση θυσία. Και το λέω αυτό διότι είναι σημαντικό σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Φώστερ και κάποιο άλλο. Για το να αναφέρονται τα επεισόδια. Ε, ε αν οι πιλότες φοβούνται νομικές συνέπειε, δεν θα αρχίσουν να πληροφορούν για επεισόδια εθελοντικά, κάτι που θα έπρεπε να κάνουν. Και εδώ τίθεται ζήτημα σε κάποια κράτη-μέλη, σε κάποιες νομοθεσίες, οι δικαστικές αρχές και αστυνομικοί μπορούν να πηγαίνουν σε τόπους ατυχημάτων και να προσπαθούν να ψάχνουν στοιχεία για την ε, δίωξη. Ε, και πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. θα πρέπει η αστυνομία να μπορεί να επεμβαίνει σε χώρους ατυχημάτων μόνο αφού έχει τελειώσει τη δουλειά της η αρμόδια ε, αρχή της πολιτικής αεροπορίας που προσπαθεί να διαρευνήσει το ατύχημα. Και εκείνη που προσπαθούν να διασώσουν τους ανθρώπους πρέπει να είναι πρώτοι και όχι οι αστυνομικέ αρχές που ψάχνουν να βρουν ποιον θα κυνηγήσουν μετά. Αυτοί πρέπει να περιμένουν μέχρι να φύγουν οι αρμόδιοι για την έρευνα των αεροπορικών ατυχημάτων από τον τόπο του ατυχήματος. Ενοχλούμε, εκνευρίζομαι με αυτό, ξέρετε. Διότι τι συμβαίνει. Αρχίζει η αστυνομία να πηγαίνει εκεί πέρα, να ερευνά και εμποδίζει τους αρμοδίους τη πολιτική αεροπορία από τη σωστή διερεύνηση του ατυχήματο. Πρέπει να προσεγγίσουμε με συμπάθεια τα θύματα και τους συγγενεί, αλλά να πετύχουμε και ισορροπία όσον αφορά και τη ρεαλιστική προσέγγιση. Πώ θα το πετύχουμε αυτό. Να ξέρουν όλοι τα πάντα σε, σε μια ώρα, υπέροχο στόχο. Εντάξει, να το προσπαθήσουμε. Είναι ρεαλιστικό στόχο. Καλύτερα να πούμε δύο ώρε και να δουλέψει, αντί να λέμε θέλουμε να ξέρουμε σε μια ώρα και να μην δουλέψει ποτέ αυτό το σύστημα. Να είμαστε ρεαλιστέ. Τροφή προσκέψη, ναι. Τέλο. Κάτι που είπαν κι άλλοι. Χρειάζεται σαφή ανεξαρτησία των ερευνητικών φορέων. Οι ερευνητέ από τους ρυθμιστές να είναι διαχωρισμένοι. Οι ρυθμιστές, οι ρυθμιστικέ αρχές δεν θα πρέπει να ανακατεύονται στην έρευνα και οι ερευνητέ δεν θα πρέπει να ανακατεύονται στη δουλειά των ρυθμιστικών αρχών. Είναι διακριτή ρόλη. Παράρτημα 13 αναφέρει η κυρία Ντεβερέκα το σύστημα και το σύστημα δουλεύει πολύ καλά. Άρα γιατί να το εξετάζουμε και να θέλουμε να το αλλάξουμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα η ΕΑΣΑ να ενταχθεί στο παράρτημα 13. Έχω όμως σοβαρό, σοβαρό πρόβλημα αν η ΕΑΣΑ εμπλακεί στις έρευνες. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζίμποντ το λόγο σε λίγο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και λέω ότι πολλά μέλη ανησυχούν. Γιατί πράγμα ανησυχούν. Ποιο θα είναι ο πραγματικό ρόλο τη ΕΙΑΣΑ. Θέλουμε από εσά 100% διαβεβαίωση ότι η ΕΙΑΣΑ δεν θα αναμειγνύεται στα τυχήματα. Λοιπόν, ο κ. Σέιμπορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω για το θέμα που αναφέρατε στο τέλος σας. Αλλά πρώτα θα ήθελα να πω ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια. Πάρα πολύ καλή η έκθεσή της. Είναι πολύ περίπλοκο θέμα και πάρα πολύ σημαντικό. Το είπαν όλοι όσοι μίλησαν. Εντυπωσιάστηκα από την ποιότητα της εκθέσεως. Είναι σημαντικό βήμα για την όλη νομοθετική διαδικασία. Και είναι κάτι που αφορά τις εργασίες της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να αναφερθώ σε κάποιους στόχους που κρύβονται πίσω από τις προτάσεις για κάποιες βασικές αρχές και κάποιες ε, όρους ε, πλαίσια που θα πρέπει να έχουμε υπόψη και να εστιαστούμε από αυτών, επί των αρχών αυτών. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει σαν στόχο να χρησιμοποιούμε καλύτερα την τεχνογνωσία και τους πόρους που έχουμε στην Ευρώπη και είναι διαθέσιμοι για την εξέταση. Λοιπόν, η πρόταση επίσης έχει και ένα στόχο την ενίσχυση του, των δυνατοτήτων που έχει ερευνητικό μηχανισμός για να χορηγεί πληροφορίες που βοηθούν την πρόληψη των ατυχημάτων. Και αυτό είναι σημαντικό και είναι τροφή προσκέψη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως ε, πολλοί είπαν ότι θέλουμε να διαφυλάξουμε και να βελτιώσουμε την προστασία των συμφερόντων των οικογενειών των θυμάτων και επίσης θεωρήσαμε κάτι που ήδη αναγνωρίστηκε κατά τις συζητήσεις ότι κάποιες διευκρινήσεις για τη διαδικασία διερευνήσεω των τυχημάτων χρειάζεται και συσχετισμό με τι άλλε διαδικασίε ποιο είναι, είναι κάτι που απαιτείται και είναι ακαθόδε, πάρα πολύ ακαθόδε θέμα για κάποια κρατημέλη. Θα ήθελα τώρα να εστιαστώ σε κάποιου τομεί ιδιαίτερης ανησυχίας. Δεν θέλω να σας αποκρύψω ότι αυτές οι ανησυχίες επίσης υπάρχουν και δημιουργούνται λόγω της θέσεως του Συμβουλίου για κάποιες από τις πτυχές. Λοιπόν, η χρήση στοιχείων διαφόρων συμβάντων. Έχουμε κάποια μέσα στη διάθεσή μας, αλλά πιστεύουμε ότι αυτές οι πληροφορίες που συλλέγονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο όπου αποτίθενται τα συμβάντα δεν χρειάζεται με αποτελεσματικό τρόπο. Το καταλαβαίνουμε. Και γι' αυτό χρειάζεται τυποποίηση των στοιχείων που διατίθεται και να διευρυνθούν ποιε δυνατότητε υπάρχουν και διευκρινιστούν οι όροι προσβάσεω στη βάση δεδομένων. Και τι άλλο συζητήθηκε και στο Συμβούλιο, ξεχωριστό κατά πόσο δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να σε αυτό το θέμα. Αν αυτό θεωρηθεί ξεχωριστό, θα καθυστερήσει κάποια βελτίωση. Καλωσορίζουμε και υποστηρίζουμε την πρόταση της εισηγήτριας για να επιληθεί το θέμα και η Άσα να είναι αρχή υπεύθυνη για τακτική ανάλυση των πληροφοριών που προέρχονται από το κεντρικό αποθετήριο αυτό συλλογή των πληροφοριών για τα συμβάντα. Των ευρωπαϊκών δίκτυων τώρα, ερευνητικών αρχών και δυνατότητες και αναγκαιότητα να ενισχυθεί το δίκτυο. Πράγματι, Πρόεδρε, αναλύσαμε, συντάσσοντας την πρότασή μας, τα θεσμικά ζητήματα. Χρειάζεται και ενδεδειγμένο δημιουργηθεί ένας νέος θεσμός για να το κάνει αυτό. Κάποιοι συνάδελφοι, κάποια μέλη Τη Επιτροπής αναφερθήκαν στο Αμερικανικό σύστημα. Αυτό είναι συγκεκριμένο στέρεο, ανεξάρτητο, είναι μια αρχή ανεξάρτητη, κάτι που δεν προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς ακολουθούμε πιο ρεαλιστικό τρόπο, βασιζόμενοι στα υπάρχοντα και διερευνώντας δυνατότητες να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους, να διαθέσουμε του πόρου με το σωστό τρόπο, διότι γνωρίζουμε αυτά που μας λένε για τα ατυχήματα ότι κάποιε χώρε είναι καλύτερα εξοπλισμένε από άλλε και πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο μοίρασμα των πόρων. Κάτι που θα βοηθούσε να εντοπίσουμε του λόγου για τα ατυχήματα ταχύτερα, αποτελεσματικότερα. Εδώ έχουμε προστιθέμενη αξία. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνει υπόψη κάποιες επιφυλάξεις που πάντα υπάρχουν όταν κάποιος προτείνει ένα νέο θεσμό, κάποιο νέο σύστημα που δημιουργεί ερωτηματικά, νομίζω ότι μπορούμε να οικοδομηθούμε σε αυτά που υπάρχουν και να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους για να ενισχύσουμε το δίκτυο αυτό, έχοντας κάποια συμπληρωματικά στοιχεία, όπως δημιουργία προγράμματος εργασίας, που ίσως θα μπορούσε να υποστηριχθεί από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ούτως ώστε να έχουμε και διάλογο μαζί σας με την Επιτροπή σας που ενδιαφέρεστε για την παγίωση του έργου για τη διερεύνηση των ατυχημάτων. Τέλος, ο ρόλος της ΕΙΑΣΑ πρόεδρε, θέσατε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων, ενδεχόμενη σύγκρουση που υπάρχει σε αυτό το τομέα μεταξύ προσεγγίσεων. Και είπατε, και λέω, δε, θα πρέπει να αναγνήσουμε τις ρυθμιστικέ αρμοδιότητες και τι ερευνητικέ τι αυτέ. Οι έρευνε θα πρέπει να διεξάγονται ανεξάρτητα από εκείνους από, ανεξάρτητα από τις ρυθμιστικές διεργασίες. Ναι, συμφωνώ. Θα διεξαχθούν περισσότερε συζητήσει σε αυτή την Επιτροπή για το σωστό ορισμό του ρόλου της ΕΙΑΖΑ. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι Ποιο θα είναι ο ρόλος της ΕΙΑΖΑ. Δεν θα πρέπει να είναι να ερευνά τα ατυχήματα και τους λόγους για τα ατυχήματα ο ρόλο της ΕΑΣΑ δεν θα πρέπει να είναι να ξεκινά κατά κάποιο τρόπο παράλληλε έρευνε για τα ατυχημάτων. Παράλληλα με εκείνους οι οποίοι άμεσα είναι επιφορτισμένοι με αυτό το έργο, διότι διαφορετικά θα δημιουργηθούν προβλήματα, θα δημιουργηθεί σύγχυση και θολούρα. Η ανεξαρτησία των ερευνητών των ατυχημάτων θα πρέπει να προστατευθεί πάση θυσία. Όμως, και θα ήθελα εδώ να το τονίσω, Συμβαίνει τακτικά κατά τη διάρκεια ερευνών για ατύχημα να προκύπτουν ερωτηματικά όσον αφορά το σωστό ορισμό, σχεδιασμό κάποιων ρυθμιστικών πραγμάτων, όπως απαιτήσει για χορήγηση άδεια πτήσεως. Και αν μια τέτοια έρευνα ενός ατυχήματος καταδείξει ότι ίσως να υπάρχει πρόβλημα με τον τρόπο που κάποιες από τις απαιτήσει καθορίζονται, τότε είναι ουσιαστικό και σημαντικό ο ρυθμιστικός φορέας που έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει για να καθορίσει τις απαιτήσει για να χορηγηθεί άδεια πτήσεων να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον επηρεασμό των ερευνών αυτών καθεαυτών. Όμως, αν επί παραδείγματι διαφανεί από κάποια έρευνα ότι κάποια διευκρίνηση για κάποιες διαδικασίες που εφαρμόζει ο πιλότο είναι αναγκαίε, διότι υπήρξε κάποια σύγχυση σχετικά με το θέμα, τότε εκείνοι που καθορίζουν τι εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να ενημερωθούν αμελητοί. Και αυτό σαν τμήμα τη διαδικασία για την αποφυγή ατυχημάτων. Αυτή η διάσταση λοιπόν, αυτό το στοιχείο τη πρόληψη των ατυχημάτων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αναγνωρίζουμε βεβαίω, βεβαίως τις αρχές της ανεξαρτησίας της είναι η ανεξαρτησία που πρέπει να προστατευτεί. Κάποια μέλη τη Επιτροπή Μεταφορών αναφέρθηκαν στο θέμα τη προστασία των δεδομένων. Είναι επίση κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιοι έθεσαν το δάχτυλο επί του κινδύνου να έχουμε, πώς το λέμε, πώς το λέμε, στη γραφειοκρατική γλώσσα, τη στάση αυτή των πληροφοριωτών, των whistleblowers, που μπορούν να εντοπίζουν κάποια προβλήματα. Θα πρέπει αυτά να τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν κανένα δύο ερωτήσεις που θέθησαν επί εκανθοδών νομικών προβλημάτων. Θα το δώσω τώρα στη συνάδελφό μου την κυρία Κουματσιώτη που ξέρει καλύτερα αυτή τη σχέση μεταξύ της έρευνας των ατυχημάτων, της σχετικής διαδικασίας και της, των παράλληλων νομικών διαδικασιών για να καθοριστούν οι ευθύνε κλπ. Ετέθησαν κάποια ερωτηματικά και ελπίζω ότι θα μπορέσει η συνάδελφος να δώσει κάποιες διευκρινήσεις, διότι είναι καλύτερα ενήμερη από το θέμα. Και τέλος, θέλω να πω το εξής. Κάποιοι συνάδελφοι πρέπει να συνεργαστούμε, συνεργαστούμε και σε κάποια φάση όταν προχωρήσει η διαδικασία συντάξης γνωμοδοτήσεως στην Επιτροπή θα πρέπει να δούμε καλύτερα ποια είναι η θέση του Συμβουλίου σχετικά με αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη να, να προσφέρει την υποστήριξή της στις ε, συζητήσεις που θα πρέπει να λάβουν χώρα συζητήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που μέχρι τώρα το Συμβούλιο, μέχρι τώρα, επί κάποιων ζητημάτων έχει διαφορετική θέση από την έξοχη έκθεση της κυρίας Ντεβεριάκ. Όλγα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ακούστηκαν διάφορα ερωτήματα σήμερα σχετικά με την ισορροπία, τη διάδραση μεταξύ δικαστικών αρχών και ερευνητικών τι αυτόν. Άρθρο 15 της προτάσεως διευκρινίζει ότι η ερευνητική αρχή ελέγχει κάποιες πληροφορίες και ότι κάποιες πληροφορίες αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο υπό ορισμένες συγκεκριμένες συνθήκες και συγκεκριμένους σκοπούς. Επίσης διευκρινίζει πότε και υπό ποιες συνθήκες ο δικαστής θα πρέπει να αποφασίσει, να δύναται να αποφασίσει, κατά πόσο λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και τα συμφέροντα της έρευνας και το κοινό συμφέρον, οι ειδικέ πληροφορίες θα πρέπει να αποκαλυφθούν. Αλλά, ξανά, αυτό απαιτεί απόφαση δικαστική, δικαστηρίο. Άρα, ο άρχοντας του παιχνιδιού παραμένει ο ανεξάρτητος ερευνητής του ατυχήματο. Και το ότι αυτή η πρόταση διατηρεί αυτά που λέει το παράρτημα 13 της συμβάσεως του Σικάγου, δηλαδή την ανεξαρτησία της ερευνητικής αρχής που ερευνά το ατύχημα, υπενθυμίζεται στο άρθρο 5 και θα δείτε τρεις διαφορετικές παραγράφους που το επαναλαμβάνουν τώρα σχετικά το ερώτημα που ετέθη, μας ετέθη από το αξιότιμο μέλο τον κύριο Φλάκαν. Δηλαδή, τη συμμετοχή του κράτου σχεδιασμού και το ρόλο του ΕΙΑΣΑ, θα ήθελα να υπενθυμίσω στην Επιτροπή ότι η ΚΑΟ αναγνωρίζει ότι τα κράτη ίσως να έχουν διαφορετικά συμφέροντα στην έρευνα. Και γι' αυτό το λόγο προβλέπεται ότι τα κράτη έχουν το δικαίωμα να διορίσουν πιστοποιημένο εκπρόσωπο, διαπιστευμένο εκπρόσωπο. Και η χώρα, όπως αναφέρεται στο παράδειγμα 13, τι λέει το άρθρο 10. Λέει το άρθρο 10 ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού για τη διασχεδιασμό τύπου του εξοπλισμού είναι εκείνος ο οποίος θα αποφασίσει και θα καθορίσει πού και ποιο κράτος μέλος θα διορίσει έναν διαπιστευμένο εκπρόσωπο. Η Φόκερ, παραδείγματο χάρη. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι Ολλανδική εταιρεία. Η Φόκερ, λοιπόν, εμπλέκεται σε ένα τύχημα. Η Φόκερ, λοιπόν, έχει βασική έδρα στην Ολλανδία. Οπότε, η Ολλανδία θα διορίσει έναν πιστοποιημένο εκπρόσωπο. Ποιος είναι ο ρόλος της ΙΑΣΑ. Ο ρόλος της ΙΑΣΑ είναι αυτός που περιγράφεται στο άρθρο 9 τώρα της προτάσεως. Η ΆΣΑ, όπως ήδη δηλώνεται στο άρθρο 20 του κανονισμού 216 του 2008, σχετικά με τις αρμοδιότητες ε, της υπηρεσίας, η ΆΣΑ λοιπόν θα ασκήσει το ρόλο της σαν σύμβουλος εκ μέρους της χώρας του σχεδιασμού. Και αυτό εξασφαλίζεται και στις δύο παραγράφους του άρθρου 9, όπου εκεί ρητά γίνεται διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και του ρόλου που θα δραματίσει η ΆΣΑ στις έρευνες που είτε διεξάγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είτε εκτός αυτής. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε. Κύριε Ντεβιράκ, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Εσείς και τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους που συμμετείχαν ε, ιδιαίτερα επικοδομητικά στην όλη συζήτηση. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα εδώ, αλλά πάντως θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Ζένκε, ο οποίος ορίστηκε σκιώδης πριν από μερικούς μήνες για αυτό το θέμα. Με τα γεγονότα βέβαια στην Πολωνία, προφανώς το θέμα έχει ιδιαίτερο βάρος. Οι διάφορες παρεμβάσεις αναφέρθηκαν γενικά μιλώντας κυρίως στην πρόσβαση στα ευαίσθητα δεδομένα, στο σημείο επαφής και στη στήριξη των θυμάτων. Για το πρώτο θέμα. Οι ευαίσθητες πληροφορίες είναι εκείνες που συλλέγουν ε, οι αρμόδιοι κατά τη διάρκεια της διερεύνησης. Είπατε ότι εφόσον εμπλεκόμενοι σε ένα τύχημα αρνούνται να απαντήσουν στην ε, διερεύνηση για την ασφάλεια ε, προκειμένου αυτά να φτάσουν στην δικαιοσύνη, επειδή το γεγονός αυτό, ε, τότε βέβαια διακυδεύεται η ίδια η διερεύνηση και η ασφάλεια. Δεν μπορεί ούτε η αρμόδια διερευνητική αρχή να κάνει τη δουλειά της, ε, ούτε και τα θύματα, οι τους να έχουν σωστά αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε περισσότερο τα δεδομένα. Υπάρχει αυτό και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό εμείς είπαμε ότι ό,τι έχει να κάνει με τα γεγονότα και με την ανάλυση των γεγονότων να πηγαίνουν στην δικαιοσύνη. Τα υπόλοιπα να κρυθούν απόρριτα. Τώρα το γεγονός ότι ορίζουμε ένα άτομο επαφής. Το Γραφείο Επιθεώρησης Προσωπικών Δεδομένων, Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων συμφώνησε με τις τροπολογίες μου. Η κυρία Άλβαρες νομίζω είπε ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το άτομο επαφής που ορίζει ο ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης δεν έχει την υποχρέωση να ορίσει άτομο. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν την υποχρέωση, εφόσον οριστεί τέτοιο άτομο, να το χρησιμοποιήσουν στην περίπτωση ατυχήματο. Να έρθουν με αυτό πρώτα σε επαφή. Κυρία Φώστερ και εσείς, κύριε Άλβαρος, νομίζω, στο, αναφερθήκατε στον κατάλογο των επιβατών. Και είπατε μέσα σε μια ώρα είναι δύσκολο να δοθεί ο κατάλογος επιβατών και να βάλουμε ε, μόλις αυτό είναι δυνατό. Αν όμως το αφήσουμε ανοιχτό το θέμα, μπορεί τελικά να βρεθούμε αντιμέτωποι με καταχρή, καταχρήσεις, τέλος πάντων, όχι επίτηδες, αλλά όπως έχει γίνει κατά το παρελθόν, με μεγάλες καθυστερήσεις. Γι' αυτό εγώ τι κάνω. Πήγα στο Ζάβεντεμ και εκεί κοιτάξαμε. Εντάξει, δεν πρόκειτο βέβαια για περίπτωση κρίση, αλλά είδαμε τι ήταν εφικτό και τι δεν είναι εφικτό. Και από την εμπειρία μα εκεί διαπιστώσαμε ότι είναι απόλυτα εφικτό να δοθεί ο κατάλογο των επιβατών μέσα σε μια ώρα από τη στιγμή που λαμβάνει η χώρα ένα τύχημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και οι οικογένειε των ε, θυμάτων επέμειναν πάνω σε αυτό, ότι γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουν τον κατάλογο επιβατών πολύ γρήγορα. Την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε είχαμε πει ναι, αλλά ο κατάλογος θα πρέπει να είναι και αξιόπιστος και όχι να έχουμε γρήγορα τον κατάλογο αλλά να μην είναι αξιόπιστος. Εννοείται, όμως με την τεχνολογία που διαθέτουμε σήμερα μπορούμε να έχουμε έναν αξιόπιστο κατάλογο επιβατών. Τώρα, ο κ. Φικεστάιν ε, έφυγε βέβαια, αλλά απάντησε έτσι καλώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε, για τον κύριο Λιμπεράσκη, τα ατυχήματα και τα συμβάντα που έχουμε σε ένα κατάλογο, αλλά για το οποίο δεν έγινε ποτέ τίποτα, το είπε και η Επιτροπή, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Ο οργανισμός αυτός που συγκεντρώνει τα στοιχεία, τα συγκεντρώνει, αλλά μετά δεν αναλύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό πρέπει να αποφεληθούμε από αυτή την ευκαιρία για να γίνεται η ανάλυση των ε, στοιχείων. Να αναλύονται αυτά τα συμβάντα, ώστε να αποφύγουμε καινούρια συμβάντα ή ατυχήματα. Έχω λοιπόν τις δικές μου τροπολογίες, περιμένω και τις δικές σας για να εμπλουτιστεί το κείμενο ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σωστά. Αναφερθήκατε πριν και στο, το πόλευ. Υπό το ατύχημα αυτό χάσαν τη ζωή τους πολλά άτομα, όπως ξέρουμε. καταλαβαίνετε ότι ό,τι εκθέσεις έχουμε για ατυχήματα και διερευνήσεις, το έχουμε ζητήσει και παλιότερα και η δικιά μας Επιτροπή και στην προηγούμενη θητεία, η αντίστοιχη Επιτροπή, να είναι η Γενική Διεύθυνση Β που ασχολείται. Υπάρχει λοιπόν ένα πρώτο σχέδιο τέτοιας μελέτης που αναθέσαμε στην Διεύθυνση Β. Αλλά δεν έχουμε αυτή τη μελέτη. Απλώς το θυμίζω στους ευρωβουλευτές ότι έχουμε ζητήσει τέτοια μελέτη. Κύριε Σκάτσιαν, θέλετε να σχολιάσετε κάτι. Σύντομα σας παρακαλώ, πολύ σύντομα. Ναι, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να υπενθυμίσω στην εισηγήτρια ότι ζήτησα τροπολογίες που έχουν προτείνει οι πιλότοι και οι ρυθμιστές κυκλοφορίες, ελεγκτές κυκλοφορίες. Έχετε κάποια άποψη για αυτές, τις έχω ήδη προτείνει, τις ξέρετε. Η κυρία Ντεβιράκ είναι σε θέση να απαντήσει. Α, ναι, καλώς. Αλλιώς σας περιμένουμε την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και μετά να κοιτάξουμε όλες τις τροπολογίες στο σύνολό τους. Αλλά δεν ξέρω αν η κυρία Ντεβιράκ μπορεί να σχολιάσει. Ναι. Α, νομίζω ότι η συγκήτρια προτιμάει να περιμένουμε και να σχολιάσει τις τροπολογίες αυτές όταν σχολιάσει και τις υπόλοιπες τροπολογίες, όταν δηλαδή έχει κλείσει η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Συμφωνεί. Ινές, Ινές, προσπαθώ να προχωρήσω. Άντε, τι θέλεις. Μετά από αυτό που είπε ο συνάδελφος, μπορεί να μην μπορεί να μιλήσει η συγγήτρια για τις συγκεκριμένες ε, τροπολογίες, αλλά για το τι μπορούν να κάνουν οι πιλότοι με τα συμβάντα στο οποία μπλέκονται η συγγήτρια, η κυρία Ντεβεράκ, θα μπορούσε να σχολιάσει λιγάκι κατά πόσο σκοπεύει να βάλει κάτι για την προστασία των ε, πιλότων, οι οποίοι αποτελούν πολύ σημαντική πηγή όταν διαρευνώνται ατυχήματα. Να μπορούν να συμμετέχουν να αποτελούν μέρος της αλυσίδας, αλλά να προστατεύονται συγχρόνως. Η κυρία Ντεβιράκ. Ακριβώς πρόκειται για την ισορροπία στην οποία αναφερθήκαμε πριν. Οι πιλότοι πρέπει και τα μέλη του πληρώματος πρέπει να μπορούν να δίνουν στοιχεία χωρίς να κινδυνεύουν από Μόνο έτσι θα προχωρούν οι διερευνήσεις και τα συμβέντα στα οποία εμπλέκονται δεν θα επαναλαμβάνονται. Αν δεν προστατεύονται, ε, δεν θα ανοίγουν το στόμα τους. Οπότε δεν θα μπορούμε να παίρνουμε μαθήματα από τέτοια συμβάντα. Γι' αυτό πρέπει να έχουν την ελευθερία να μιλούν, χωρίς όμως να φοβούνται ότι θα διωχθούν με κάποιο τρόπο στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, είναι σημαντικό πιστεύω και εγώ να συζητήσουμε όλες τις τροπολογίες όταν τις έχουμε είτε προέρχονται από πιλότους είτε από άλλη πλευρά και να θυμόμαστε ότι οι τροπολογίες όμως που εξετάζουμε είναι τροπολογίες ευρωβουλευτών και όχι πιλότων. Την κάνω αυτή τη διάκριση, έτσι. Προσοχή. Πάντως, 31 Μαΐου είναι η προθεσμία. Ε, Ιουνίου θα ψηφίσουμε και μετά τον Ιούλιο θα πάει το θέμα στην Ολομέλεια. Προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών των Ευρωβουλευτών είναι η 4η Μαΐου. 4 Μαΐου προθεσμία συζήτηση στις 31 Μαΐου. 1η Μαΐου ψηφίζουμε και το θέμα πάει στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. 4 Μαΐου προθεσμία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ντεβιράκ και όλους όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση. Και περνάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι η εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Can I make my usual plea that all meetings, Commission, Parliament. Όλες οι ομάδες, λόμπι ή οποιοδήποτε άλλοι είναι εδώ και συζητάνε να βγουν από την αίθουσα. Εδώ πρόκειται για συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταφορών, οπότε οι υπόλοιποι να βγουν, να πείτε και στους υπόλοιπους τι ωραία που είναι εκεί έξω. Οπότε όσοι δεν έχουν θέση εδώ να βγουν. So, the mass exodus from the room, I take it, has nothing to do with me personally. Φαντάζομαι ότι δεν είναι επειδή παρουσιάζω εγώ το θέμα που φεύγει τόσος πολλής κόσμος από την αίθουσα. Θα θυμόσαστε ότι οι συντονιστές ε, συμφώνησαν ότι ο Πρόεδρος θα έπρεπε να υποβάλει ένα ψήφισμα εκ μέρου τη Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση τη πρώτη δέσμη μέτρων για του ε, σιδηροδρόμου. Έχετε λάβει λοιπόν αυτό το ψήφισμα, το προτινόμενο ψήφισμα, το οποίο ακολουθεί την πρώτη συζήτηση που είχε γίνει τον ε, Φεβρουάριο και μετά την ε, διαβίβαση της δεύτερης έκθεσης σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των ε, εξελίξεων την οποία λάβαμε τον τελευταίο Δεκέμβριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2012 εκαπα Τώρα, μετά την εφαρμογή αυτών των μέτρων η ε, ε, μεταφορά επιβατών ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου του 2010 και το 2006 και 2007 άνοιξε, άνοιξαν τα σύνορα σε ό,τι αφορά τις, τη μεταφορά φορτίων συνδρομικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε πως αυτή η πρώτη δέσμη μέτρων ε, είχε προβλεφθεί για το Σεπτέμβριο του 2010, αλλά το νομικό και το θεσμικό πλαίσιο Υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε κάποια παράπονα σε ό,τι αφορά τη μη ε, σωστή εφαρμογή των ε, πρώτων, της πρώτης θεσμής μέτρων για τους σιδηροδρόμους με αποτέλεσμα να αποσταλούν αντίστοιχα παράπονα σε, στα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρείται πως δεν απάντησε επαρκώς ε, σε αυτές τις ε, ερωτήσεις σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και κατά συνέπεια η Επιτροπή μας αποφάσισε να συντάξει το λόγο ψήφισμα. Εγώ σε αυτό το ψήφισμα προσπαθώ να αντικατοπτρίσω τα όσα συζητήθηκαν και βέβαια να λάβω υπόψη της νόμης των συντονιστών σας. Αυτό λοιπόν που αναφέρουμε είναι η έλλειψη ανάληψη ενέργεια από πλευρά των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τη πρώτη τέσσερι μέτρων και επίση ασκεί κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τον έλεγχο από την πλευρά τη ε, απέναντι στα κράτη-μέλη, καθώ καμία ενέργεια δεν λύθη από τη δική τη πλευρά κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Άρα το ψήφισμα ε, εστιάζει σε τρία ε, ζητήματα. Πρώτον, η έλλειψη ανεξαρτησίας ενός διαχειριστή των υποδομών, η σωστή κατανομή των δυνατοτήτων στα εθνικά δίκτυα ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα πρακτικά ε, ζητήματα εφόσον αυτός ο διαχειριστής σχετίζεται με την εταιρεία εκμετάλλευσης, με την εταιρεία παροχή υπηρεσιών, μετά η έλλειψη αντίστοιχων καονιστικών μηχανισμών και αντίστοιχων αρμοδίων ε, για να επιλύουν ζητήματα ρυθμιστικά και μετά η επιβολή ε, σχετικών ε, τέλων η οποία γίνεται με τρόπο αναποτελεσματικό και αδιαφανή. Και όπως βλέπετε χρησιμοποιώ διπλωματικές εκφράσεις εδώ όταν λέω δεν είναι επαρκώς διαφανές το σύστημα αυτό. Κατά αυτόν τον τρόπο ε, υπάρχει δυσκολία για την ένταξη νέων επεκτών, νέων επιχειρήσεων σε αυτή την αγορά. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται δηλαδή είναι να ακολουθείτε μια πολιτική προστατευτισμού. Άρα λοιπόν εδώ αυτή, αυτό το ψήφισμα έρχεται να σχολιάσει την αναθεώρηση της πρώτης θέσης για του συντριοδρόμους. Όπως σας ξαναείπα, οι συντονιστέ επιθυμούσαν να συνταχθεί ένα τέτοιο ψήφισμα. Είναι το προϊόν λοιπόν αυτή τη βούλησή του. Και βέβαια θα ήθελα τώρα να ακούσω τι δικέ σα απόψει. Και ξεκινάω με τον ε, κύριο Γκρόσιο για το ΕΛΚ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω α, τον συγκητή μας καθώς κατέγραψε τα όσα είχαμε πει τόσο εδώ όσο και στο Στρασβούργο σε σχέση με αυτό το ζήτημα στην Επιτροπή μας, οι επιπτώσεις δηλαδή τη μίσος της εφαρμογής αυτών των διατάξεων ή η ασφαλμένη εφαρμογή αναφέρονται μέσα σαφήνεια μέσα σε αυτό το σχέδιο ψηφίσματος. Δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω. Ε, με βάση την εμπειρία μου, όταν λέμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να κάνει το ένα και το άλλο χωρίς να αναφέρουμε συγκεκριμένα πράγματα δεν, δεν έχει νόημα. Το να, καλύτερο θα ήταν να λέμε without, δηλαδή να λέμε without delay, δηλαδή χωρίς καθυστέρηση εκεί κάπου στο 3 μπορούμε για παράδειγμα να πούμε σε 6 μήνες. Και αυτό ισχύει ε, και για μια σειρά από ακόμα σημεία στο 4 και σε μια σειρά άλλα σημεία το 10 για παράδειγμα όπου καλύτερο θα ήταν να αναφέρουμε συγκεκριμένη προθεσμία. Δηλαδή όπου ζητάμε να μας διαβιβαστούν συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεκριμένες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και ειδικότερα στα 3, 5 και 10 καλό θα ήταν όχι μόνο να ζητάμε καλής ποιότητας δεδομένα αλλά και να θέτουμε συγκεκριμένα, συγκεκριμένη προθεσμία. Ε, ίσως ε, ε, στο 2016 ενδεχομένω θα μπορούσαμε να κάνουμε και λόγο ή όχι πάλι για το πλήρες άνοιγμα της αγοράς των συνδρομικών μεταφορών. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο. Αυτό που αφήνεται σε εσάς. Presidente, intervengo a Αντικαθιστώ τον συντονιστη Ελ Κατράουι που δεν μπορεί να είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Η ομάδα μου είναι υπέρ της πρότασης ψηφίσματος. Επιμένουμε όμως πάνω σε μία πολύ σημαντική για μας πτυχή Δηλαδή θέλουμε να ζητάμε από τα κράτη-μέλη να επενδύουν σε υποδομές. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε μια πραγματική ελευθέρωση του συνδρομικού δικτύου και να μπορέσει αυτός να είναι και ανταγωνιστικός. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αποφεληθούμε από νέες συνθήκες ανταγωνισμού για τους σιδηροδρόμους μας. Ευχαριστώ κύριος Στέρξ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ζήτησα το ψήφισμα αυτό και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να σε περιλαμβάνει τα πιο στοιχειώδη και να είναι αυτά ξεκάθαρα. Εννοείται ότι η εφαρμογή των οδηγιών, των, του πρώτου πακέτου οδηγιών, δεν έχει προχωρήσει όπως θα έπρεπε. Είναι ξεκάθαρο από το κείμενο. Οπότε, αυτό που πρέπει να ξεκαθαριστεί εδώ είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος που είναι να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή δομή για τους σιδηροδρόμους. Αυτή είναι η αρχή και αυτήν πρέπει να επαναλαμβάνουμε. Μέσα σε 20 χρόνια δυστυχώς δεν έχουμε προχωρήσει. Είμαστε πολύ πίσω, το είπατε κι εσείς. Υπάρχουν προστατευμένες αγορές. Εγώ τι ακούω από το σχετικό κλάδο. Τα σχόλιά τους είναι ότι ζητάμε όλο και περισσότερο αμοιβαιότητα. Επίγει λοιπόν να επαναλάβουμε την αρχή ότι θέλουμε μια ευρωπαϊκή αγορά σιδηροδρόμων. Αυτό πρέπει να επαναλάβουμε. Και αυτό να το ξέρει και η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να τους ρωτήσουμε τι έχουν να απαντήσουν. Γιατί δεν εφαρμόζουν τις οδηγίες. Αυτά τα πράγματα λοιπόν πρέπει να συμπεριληφθούν για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το κείμενό μας. Εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπενθυμίσουμε ότι η αρχή ήταν αυτή δεν κάνατε αυτό που έπρεπε να το κάνετε. Συμφωνώ με τους σοσιαλιστές να ερευνήσουμε το δίκτυο. Γιατί, τι πρέπει να βελτιώσουμε. Αλλά ακόμα και εκεί που έχουν γίνει επενδύσεις, εξακολουθεί να υπάρχει μια ανατροπή μονοπωλίου. Αυτή πρέπει να αλλάξει. Μόνο να αλλάξει αυτή, θα μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Γι' αυτό θα ήθελα για αυτά τα δύο σημεία να πούμε κάτι πιο έντονο στο κείμενο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κράμερ, εκ των Πρασίνων. Ε, το ψήφισμα αυτό βασικά δεν χρειάζεται. Ή δεν θα χρειαζόταν εάν η Επιτροπή είχε ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και είχε αναλάβει δράση όπου χρειαζόταν. Εάν είχε κάνει όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε δεν θα χρειαζόταν μετά από τόσα χρόνια να προβαίνουμε σε ένα ψήφισμα. Πραγματικά δηλαδή δεν είναι απαράδεκτο το 2001 να έχουν αποφασίσει από κοινού τα θεσμικά όργανα, έτσι, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι. Ε, τα κράτη-μέλη όλα αυτά είχαν συμφωνήσει από τη δική τους πλευρά. Έπρεπε λοιπόν η εφαρμογή να είχε λάβει η χώρα το 2003 και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένει πέντε χρόνια μέχρι να κάνει κάτι. Γιατί κουνάτε το κεφάλι, αφού δεν κάνατε, γιατί δεν κάνατε τίποτα. Γιατί δεν κάνετε τίποτα. Γιατί δεν προσφύγατε στο δικαστήριο όταν είδατε ότι τα κράτη-μέλη δεν κάνουν τίποτα. Γιατί δεν κάνατε μια ε, ε, ενημερωτική εκστρατεία. Εμεί θα σα υποστηρίζουμε από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Δεν κάνετε τίποτα. Εξακολουθείτε να μην κάνετε τίποτα και τώρα εμεί τι κάνουμε. Δηλαδή, σα παρακαλάμε με ένα τέτοιο ψήφισμα να αναλάβετε δράση. Πραγματικά είναι ευγενική αν θέλετε δική μα κίνηση, αλλά αποτελεί κόλαφο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν ανταποκρίθηκε στι υποχρεώσει τη. Γι' αυτό πληρώνεται, αλλά δεν έπραξε αυτά που πρέπει να πράξει. Από εκεί και μετά. Ε, εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε αυτέ τι μεταρρυθμίσει στην αγορά των συνδημοτικών μεταφορών είναι να υπάρχει περισσότερο ανταγωνισμό. Αλλά αν δούμε με πόση ε, πόσο αγνοούνται οι διάφορες ε, πραγματικά αθέμητες πρακτικές οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν πραγματικά έχουμε, μας δημιουργείται τεράστια έκπληξη. Μιλάμε, μιλάμε λοιπόν για έχουμε μια, μια ανταγωνιστική αγορά που έχει πολύ ψηλέ ε, τιμέ. Ε, και ε, πραγματικά αυτό το επιτρέπουν. Το επιτρέπουν τα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, στη Σλοβακία έχουμε τα υψηλότερα δυνατά τέλη στι συνδρομητικέ μεταφορέ. Αλλά όχι στι οδικέ του μεταφορέ. Και σα λέω για ένα ποσό το οποίο διπλάσιο, για παράδειγμα, από ό,τι στη Γερμανία. Δηλαδή, μα λέτε ότι θα πρέπει η κυκλοφορία να, να πάει σε άλλου οδούς σε άλλε οδού μεταφοράς, θα πρέπει να κάνουμε κάτι, αλλά τελικά τίποτα δεν συμβαίνει. Το ίδιο δεν συμβαίνει και στις αερομεταφορές, ε, φορητή ροζίνη ε, και ούτω καθεξής. Και το ίδιο συμβαίνει κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τα καύσιμα των ε, αμαξοστοιχειών. Και τι λέμε, ότι από το 2012 με την απελευθέρωση των αγορών ε, θα, και η ηλεκτρική τροφοδοσία των ε, σιδηροδρόμων ε, θα πρέπει να διατεθεί, να ιδιωτικοποιηθεί δηλαδή. Σας παρακαλώ, όταν σκεφτόμαστε όλα αυτά, να, σκεφτείτε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα όλε αυτέ τις προποθέσει και να δούμε τι συμβαίνει εδώ. Και γι' αυτό δεν μ' αρέσει και στο ψήφισμα. Δηλαδή θα πρέπει να πούμε καταρχήν έχουμε έναν αθέμητο ανταγωνισμό, έχουμε μια κατάσταση απαράδεκτη αυτή τη στιγμή η οποία έρχεται σε διαμετρική αντίθεση με του στόχου μα. Ένα ε, κλάδος ο οποίο λειτουργεί σωστά όχι μόνο επειδή ευθύνεται για ένα μεγάλο ποσοστό των εκπομπών στην Ευρώπη, αλλά και επειδή έχουμε αύξηση των σχετικών τιμών παρότι έχουν επενδυθεί σε αυτά τα δίκτυα δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στις τελευταίες δεκαετίες. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο πραγματικά ανταμείβει εκείνους οι οποίοι ρηπαίνουν περισσότερο και προστατεύει όσους, ε, ανταμείβει όσους ρηπαίνουν περισσότερο και έχει κυρώσεις για όσους ρηπαίνουν λιγότερο. Θα πρέπει να αλλάξουμε αυτό το σύστημα. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, και εγώ ε, για την ε, σύνταξη αυτού του ψηφίσματος. Όπως είπαμε και στην συνεδρίαση των συντονιστών, δεν διαπιστώνουμε ή δεν θεωρούμε πως μπορεί με αυτή την πρώτη δέσμη μέτρο να ισχύσει μία λύση ενιαία για όλους. Τα όσα είχαν συμφωνηθεί το 2001 δεν είχαν ακόμα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά από τα σημερινά κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε κάποιες ιστορικού και γεωγραφικού χαρακτήρα ε, διαφορές προτού κατηγορήσουμε ορισμένες ε, χώρες ε, για την μη εφαρμογή. Για παράδειγμα, η Φιλανδία και κάποιε χώρε τη Βαλτική. Εντάξει, δεν ξέρω τόσο καλά για τη Φιλανδία, αλλά οι χώρε τη Βαλτική, σα λέω, έχουν ε, ένα ε, ψηλό ποσοστό ε, συνδιοκτησία σε ό,τι αφορά τα συνδρομικά δίκτυα, γύρω στο 50%. Και χάνουμε αυτό το ποσοστό λόγω της ανάγκης εφαρμογής αυτού του, αυτής της δέσμης μέτρων. Ε, και αν δεν είχαμε συγχρηματοδότηση, δηλαδή ενισχύσει ε, κρατικές, ε, δεν θα ήταν δυνατόν να επιβιώσει αυτός ο τομέας. Ακόμα σας λέω και για τι κρατικές επιχειρήσεις δεν θα ήταν βιώσιμες. Συχνά οι, οι μεταφορές αυτές ξεκινάνε από τις χώρες ΕΑΕΣ, Ρωσία και λοιπές και φτάνουν στα δικά μας λιμάνια. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα συνολικά τέλη που θα πρέπει να καταβάλει κανείς, ε, δηλαδή ως μεταφορική εταιρεία για την ε, μεταβίβαση ενός ε, φορτίου. Στην περίπτωση της Λετωνίας, για παράδειγμα, έχουμε τρεις operators εδώ. Δύο από τους οποίους βρίσκονται στους Σολυμένα και ο ένας από αυτούς ανήκει, είναι κρατικός. Οπότε, αν έχουν αυτοί οι δύο διαφορετικές ε, τιμές, μιλάμε για ένα είδος αθέμη του ανταγωνισμού. Στη δική μας λοιπόν ε, περίπτωση δεν τίθεται θέμα ανταγωνισμού των ε, σιδηροδρομικών μεταφορών σε σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη, αλλά μιλάμε για ζητήματα ανταγωνισμού με τρίτες χώρες. Άρα λοιπόν, όταν λέμε ότι ε, προτείνουμε αναθεώρηση τη πρώτη μέση μέτρων για του σιδηροδρόμου το 2010, ίσω θα πρέπει να προσθέσουμε και να πούμε ότι λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών, ιστορικών και ούτω καθεξή ιδιαιτεροτήτων των κρατών Γιατί σας λέω ότι εάν προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε μια τέτοια ενιαία λύση, τότε πραγματικά το δικό μας το ποσοστό θα μειωθεί ακόμα

Σχετικά με το ψήφισμα αυτό για το πρώτο πακέτο οδηγιών, θέλω να επιστήσω την προσοχή σα πάνω σε μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα στο πακέτο αυτό καθ' αυτό. Θα θυμόσαστε ότι πρόκειται για ένα πακέτο οδηγιών. Και πρόκειται για την εφαρμογή τους, η οποία απαιτεί κάποια ελαστικότητα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Η αξιολόγηση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, βασίζεται στο λεγόμενο soft law που επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες. Στη μη δεσμευτική νομοθεσία δηλαδή. Για ορισμένες χώρες οι σιδηρόδρομοι λειτουργούν κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Μην ξεχνάμε ότι το πρώτο πακέτο ετοιμάστηκε το 2001. και είχε να κάνει με τις συνδρομικές αγορές των τότε 15 χωρών μελών. Η κατάσταση στις νέες χώρες μέλη είναι τελώς διαφορετική. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν πρόκειται για τις οικονομικές πτυχές του πακέτου. Επενδύσεις, διαχείριση, ε, χρέη. Αν λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, πρέπει να επικεντρωθούμε στην ε, διαφύλαξη ενός ίδιου επίπεδου για όλους. Θέλουμε επίσης να έχουμε και την εγγύηση για σωστές ε, επενδύσεις. Οπότε, εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά πιστεύει ότι είναι σωστά τα επιχειρήματα, γιατί περίμεναν τόσα πολλά χρόνια προκειμένου να φροντίσουν για την εφαρμογή του πρώτου πακέτου, ο κύριος Λιμπεράσκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Στην Ευρώπη Δέκα μέρες δεν μπορούσαμε να πετάξουμε. Δεν μπορέσαμε να έχουμε κανονικά την ολομέλειά μας στο Στρασβούργο. Και αυτό οφείλεται σε ένα πρόβλημα μεταφορών. Πρέπει να αλλάξουμε τη στάση μας λοιπόν. Και να έχουμε δύο πανευρωπαϊκά συστήματα για να ταξιδεύουμε. Το ένα να βασίζεται στην αεροπορία και το άλλο στους σιδηροδρόμους. Όταν υθετήσαμε το πακέτο αυτό το 2001, πηγαίναμε Βρυξέλλες, ε, Βαρσοβία σε 16 ώρες κατευθείαν. Τώρα τα τελευταία 4 χρόνια δεν είναι πλέον εφικτό κάτι τέτοιο. Και αυτό οφείλεται στην ελευθέρωση των σιδηροδρόμων. Είμαστε σήμερα σε μια κατάσταση όπου σε ορισμένες χώρες οι επενδύσεις για τη συντήρηση των υποδομών και για την διαχείριση είναι 4.000 το χρόνο ένα χιλιόμετρο. Αλλού 130 ή 400.000 ευρώ. Εκτιμώ λοιπόν πολύ το γεγονός ότι η έκθεση εκπονήθηκε και υπάρχουν τρεις τομείς τους οποίους τόνισε ο πρόεδρος και τα σημεία 3, 5 και 10 τα οποία ανέφεραν οι συνάδελφοι. Η κατάσταση έχει ως εξής. Οι κυβερνήσεις ακούν τους φορείς που δρούν στους σιδηροδρόμους και η Επιτροπή ακούει τις κυβερνήσεις. Αν δείτε ποια κράτη τήρησαν και φάρμοσαν τις ε, οδηγίες του πρώτου πακέτου, είναι μόνο η Μάλτα και η Κύπρος που δεν έχουν σιδηροδρόμους. Αναφέρεται και η Ιρλανδία και η Φιλανδία και η Βουλγαρία. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό. Τέλος, πρόεδρε, στο σημείο 14, όπου μιλάμε για ελλειπείς ε, επενδύσεις όσον αφορά τις υποδομές, θα έπρεπε να αναφέρουμε και την επιθυμία μας να εφαρμόσουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο σιδηροδρόμων. Όπως έχουμε με τους ευρωπαϊκούς εφαίρες. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φρομήσει και για ενία τέλη στις υποδομές στη Σουηδία. Είναι 30 cents, 6,5 ευρώ στην Πολωνία, στη Γερμανία 2 και μισό ευρώ. Πώς λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε για έναν ευρωπαϊκό χώρο σιδηροδρόμων στην... εδώ. Δεν υπάρχει. Ίσως θα έπρεπε να το αναφέρουμε αυτό. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ τον Πρόεδρο για την πρωτοβουλία που ανέλαβε και για το ψήφισμα αυτό, το οποίο ελπίζω να βοηθήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριος Κούν. Thank you, Mr. Chairman. Auch, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Σίμψον, ε, για το γεγονό ότι με, ε, με αυτό το σχέδιο ψηφίσματο θα προσπαθούμε να ασκήσουμε περισσότερε πιέσει, ούτω ώστε η μεταρρύθμιση των αγορών σε να προωθηθεί και το πακέτο μέτρων να εφαρμοστεί σωστά. Ε, το ζητούμενο είναι ότι τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία επέτρεψαν την απελευθέρωση των δικών τους αγορών είδαν να αυξάνονται πράγματι και ο κλάδος των μεταφορών και ο κλάδος της μεταφοράς επιβατών. Και ίσως καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει ποιες ακριβώς ήταν εξελίξεις στα ε, επιμέρους κράτη-μέλη, ως προς το πώς εξελίχθηκε δηλαδή ε, κλάδος της μεταφοράς φορτίων και απεβατών. Αυτό θα μας έδειχνε πού λειτουργήσε καλά, αν θέλετε, η εφαρμογή του πρώτου πακέτου και πού όχι. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και τις 21 διαδικασίες παραβάση που έχουν ε, εγκινηθεί κατά κρατών μελών. Υπάρχουν ταυτόχρονα και, κάποια, και κάποιες σαφείς καταστάσεις, ε, ε, δηλαδή το σίγουρα η σχετική διαδικασία για το Ηνωμένο Βασίλειο αφορά και την ιδιωτικοποίηση, ενώ ε, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κατά της Γερμανίας υπάρχει εδώ μια εταιρεία holding που έχει αναλάβει το 100%. Και τέλος έχουμε και κάποια άλλα κράτη-μέλη τα οποία έχουν ε, χρησιμοποιούν διαφορετικούς μηχανισμούς ώστε να έχουν το σωστό διαχωρισμό εκείνο ε, που θα πρέπει να υπάρχει είναι μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή όπως υπάρχει και στη Γερμανία σε όλα τα κράτη-μέλη, η οποία έχει άμεση αρμοδιότητα ε, όλοι οι operators οι οποίοι ε, έχουν ανάγκη δρομολόγια να μπορούν να το λαμβάνουν. και το μερίδιο αγορά των ξένων επιχειρήσεων βρίσκεται στο 23% σε ό,τι αφορά τη μεταφορά επιβατών και σε ό,τι αφορά τη μεταφορά φορτίων στο 20%. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι σχετικέ διαδικασίε ε, κατά παράβαση που κινούνται να κινούνται λαμβάνοντα υπόψη και αυτά τα ζητήματα. Και σα ξαναλέω, α μα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ εξελίχθηκε η κατάσταση, πώ αναπτύχθηκε η αγορά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ε, πέντε ετών στα διάφορα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για αυτή την πρόταση ψηφίσματος. Πιστεύω ότι αν μη τι άλλο εντοπίζει τα προβλήματα που συζητάμε κατά τα άλλα σε θέματα όπως εκείνο του κυρίου Μαρινέσκου. Σχετικά με το σημείο 7 που μιλάμε για την έλλειψη νομικών εγγύσεων θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα πρόσφατο συμβάν αρχές της χρονιάς όπου ένας φορέας όπου ήθελε να εξυπηρετήσει τη διαδρομή Μιλάνο-Παρίσι τα έχει όλα ετοιμάσει από ό,τι λέει και τις παραμονές της έναρξης παροχής αυτής της υπηρεσίας, απορρίφθηκε η γραμμή αυτή, γιατί κάτι έλειπε, πιστοποίηση, δεν ξέρω κάτι. Είναι ένα σημαντικό συμβάν. Θέλω να ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε ξέρει τι έγινε. Έχει άποψη για το θέμα. Θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και κάτι γι' αυτό, μια σύσταση, να μην ξανασυμβεί το ίδιο. Ότι δηλαδή η έλλειψη εγγύσεων οδηγεί έναν φορέα ο οποίος είναι έτοιμος καθόλου μια εβδομάδα πριν αρχίσει να λειτουργεί η γραμμή εισπράττει το όχι από δεν ξέρω ποιον. Δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός ο οποίος εμπόδισε την έναρξη της παροχής αυτής υπηρεσιών. Η κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ για το ψήφισμα. Έχω διάφορα σχόλια. Καταρχήν, θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή θα μπορούσαμε να έχουμε μια σαφή διάγνωση γιατί τα κράτη-μέλη δεν έχουν εφαρμόσει το πρώτο ε, συνδρομικό πακέτο. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω, οι άλλοι μπορεί να ξέρουν περισσότερα ή να έχουν μελετήσει περισσότερο το θέμα. Εγώ πάντως έχω την εντύπωση ότι πάντα αποφασίζουμε χωρίς να ξέρουμε. Μπορούμε να έχουμε τη διάγνωση. Γιατί? Για να μπορέσουμε να πάρουμε και τις κατάλληλες αποφάσεις. Σχετικά με το γιατί Όλα αυτά τα χρόνια τόσες χώρες δεν έχουν θέσει εφαρμογή το πρώτο πακέτο οδηγιών. Στο σημείο 2 αναφέρονται οι χώρες που δεν έχουν ε, εφαρμόσει και είναι η Γερμανία, Δανία, Εστονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθανία, Λουξεμβούργο κλπ. κλπ. Δηλαδή Άλλε χώρε. Δεν αναφέρεται εδώ η Λετωνία, λέει ο Μιλήτρια. Δεύτερον, στο, στην Ευρώπη δεν κάνουμε τα πράγματα σοβαρά για τις μεταφορές. Γιατί αν από το 2001 έχουν περάσει τόσα χρόνια χωρίς να έχουν εφαρμοστεί οι οδηγίες αυτές, συζητάμε στο Κοινοβούλιο πώς θα δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο δρόμων. τι νόημα έχει. Μα ελέγχει κανείς για όλα αυτά τα μέτρα, πέρα από τη μη εφαρμογή του πρώτου πακέτου, ελέγχει κανείς τι γίνεται με τις κατά προτεραιότητα γραμμές που έχουμε ορίσει στην Ευρώπη. Έχουμε καμιά διάγνωση γιατί δεν εφαρμόζονται αυτά που θα έπρεπε να εφαρμόζονται, τι ευθύνε έχουν τα κράτη-μέλη. Εμείς εδώ από την Ευρώπη δεν πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία εμένα με εκπλήσουν στην πολιτική της Ευρώπης. Εγώ είμαι καινούργια εδώ και εκπλήσωμαι πάρα πολύ. Τέλος το είπε και κάποιος άλλος. Ε, εμείς που είμαστε πολιτικά υπεύθυνοι και πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνε μας, ε, δεν το κάνουμε. Δεν αναπτύσσουμε τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ενώ κάθε μέρα σε όλες τις συζητήσεις, σε όλα μας τα ψηφίσματα, μιλάμε για την προστασία του περιβάλλοντος, για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που πρέπει να μειωθούν. Μα δεν είμαστε σοβαροί με τη δουλειά που κάνουμε. Ας σοβαρευτούμε. Μπορεί να χρειάζονται χρήματα. Να έχουμε περισσότερες επενδύσεις. Ναι, αλλά α έχουμε αν μη τι άλλο ένα ξεκάθαρο σχέδιο για να το πετύχουμε αυτό. Είναι οι επενδύσει που λείπουν, είναι κάτι άλλο. Τι φταίει. Εγώ πιστεύω ότι η κρίση από την οποία περάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την έκρηξη του ηφαιστείου και η συζήτηση που έγινε υπό Ισπανική Προεδρία με τον Επίτροπο Μεταφορών κατέδειξε ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε αρκετό συντονισμό και πάνω απ' όλα ότι πρέπει να δημιουργήσουμε και να αναπτύξουμε την διαλειτουργικότητα. Με αυτό τον τρόπο που πάμε τώρα δεν πάμε στο σωστό δρόμο. Και το ψήφισμα αυτό δεν θα λύσει τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος ο κύριος Κάντσεν. Ehm, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω, ακούγοντας και τους προλαλήσαντες, ότι χρειάζεται να κάνουμε διάξη κατά την την υποδομή και την κίνηση, αν θέλετε. Νομίζω ότι το πακέτο πάει προς τη δεύτερη κατεύθυνση, δηλαδή τη λειτουργία, την κίνηση την κινητοποίηση. Αν σταματήσουμε στη υποδομή, θα πρέπει να συντονιστούμε και με τα διευρωπαϊκά δίκτυα ε, όσον αφορά τον προγραμματισμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ έχουμε τη μεταφορά επιβατών, έχουμε τα τρένα υψηλή ταχύτητα, μεγάλη δυναμικότητα, ε, μεταφορά εμπορευμάτων. Ε, χρειάζεται εξορθολογισμό στι συνδρομικέ μεταφορέ, χωρί να λάβουμε υπόψη και τις άλλες μορφές μεταφορών. Αυτά θα τα δούμε στην ανα... μεταρρύθμιση των δικτύων των διευρωπαϊκών. Μετά θα δούμε και τη χρηματοδότηση όσον αφορά τι υποδομέ. Ε, εκεί θα πρέπει να πάμε προς την οθέτηση και ενίσχυση ε, των διαφόρων μέσων. Η σημασία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Το σημερινό μας θέμα είναι ότι πρέπει να διαφυλάξουμε την απελευθέρωση της αγοράς. Αν θέλουμε να έχουμε ελεύθερη αγορά, λοιπόν, με ισότιμες συνθήκες για όλους, με τους ίδιους κανόνες και τις ίδιες συνθήκες, πιστεύω, αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα επιλύσουμε το ζήτημα. Αυτό που λείπει βλέποντας το ψήφισμα στα 10 Ιουλίου του 2007, βλέπουμε το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη αυτά που θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη έκαναν ό,τι ήθελαν. Και αυτό είναι μια κοροϊδία και είναι ανύπαρκτος έλεγχος. Θα πρέπει η έκθεση να βασιστεί κατά πάρα πολύ στην ελεύθερη αγορά, σε έναν επαρκή έλεγχο για να φτάσουμε σε μια αγορά που είναι πραγματικά ελεύθερη, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ε, ισότιμη, μια σωστή απάντηση, αντίστοιχη απάντηση που απαιτείται στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Ευχαριστώ. Μάικλ, ήθελες να πεις κάτι σε απάντηση όσον είπε και ο Ζήλερ. Ε? Ναι, προέκυψαν κάποια ερωτήματα. Καταρχήν, γιατί είναι τόσο δύσκολη η εφαρμογή. Ο της ε, Ντόι Σεπάν είχε πει κάποτε ότι εκείνος ο οποίος ελέγχει το δίκτυο θέλει να είναι ο αρχηγός, ας το πούμε έτσι, ο άρχοντας. Και αυτό συμβαίνει πάντοτε, δηλαδή οι κυβερνήσεις δεν επιθυμούν να ανοίξουν πραγματικά τις αγορές ε, ε, ακολουθούν δηλαδή τις οδηγίες που τους δίνουν οι δικές τους, η δική τους εθνική επιχείρηση και ε, κατά συνέπεια δεν σημαίνει τίποτα. Δεν, δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι καινούριο. Μετά, εκείνο που λέμε είναι τα χρήματα. Κάναμε και μια ανάλυση εδώ. Δηλαδή, πού πάνε αυτά τα χρήματα. 60% ε, πάνε στις οδικές μεταφορές, πάνε στους αυτοκινητόδρομους, το 20% πάει στους σιδηροδρόμους. Αλλά είχαμε πει εμείς και προηγουμένως ότι θέλαμε 40% για τους σιδηροδρόμους. Ο κύριος Μπαρό τότε από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν υπέρ αυτή τη πρωτοβουλία, αλλά τα κράτη-μέλη ήταν κατά. Λάβετε όμω και εσεί κάποιε πρωτοβουλίε ώστε να κατευθυνθούν προ τι ε, ε, σωστέ μεταφορέ σωστές τα ε, κονδύλια αυτά. Στο ψήφισμα τώρα του 2007 λέγαμε και κάτι ακόμα. Όταν τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία είχαν απελευθερώσει τι αγορέ, για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 60%, οι κάτω χώρε συν 40%, η Πολωνία συν 30%, η Γερμανία συν 20%. Αυτέ ήταν αυξήσει στον τομέα των μεταφορών. Ενώ αντίθετα οι χώρε οι οποίε ακολούθησαν προστατευτική πολιτική όπω η Γαλλία σημείωσε συρρήκνωση του τομέα κατά 28%. Άρα λοιπόν μας, ε, μας αναφέρεται ξανά και ξανά ότι η λειτουργία και, η ίδια, και τα ίδια τα δίκτυα δεν μπορούν να διαχωριστούν στους σιδηροδρόμους. Αλλά αυτό μας το λένε επανειλημμένα κάποιοι παρότι έχουμε δει ότι αυτό ισχύει. Ισχύει δηλαδή τα δίκτυα έχουν διαχωριστεί από, τις, ε, από τη λειτουργία. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ένα απελευθερωμένο ε, τομέα. Σε ό,τι αφορά αυτή την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέτυχε ε, και γι' αυτό είναι μια καλή πρωτοβουλία αυτό το ψήφισμα. Μόνο γι' αυτό ε, πήρα το λόγο, για να δώσω αυτέ τι απαντήσει, Πρόεδρε, Ευχαριστώ πολύ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριο Καστελότη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριο Καστελέτη. Καστελέτη. Κύριε Καστελέτη, θα πρέπει να ξεκινήσετε τη δικασία παράβαση παράβασης εναντίον μου. Θα περιμένω την επιστολή σας σε, σε μια δεκαετία. Κύριε Καστελέτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Εν γέννη, νομίζω ότι το ψήφισμα ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση, αλλά καμιά φορά κανείς υπεραπλουστεύει και να εξηγήσω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε αιτιολογημένη γνωμοδότηση τον Οκτώβριο, 8 Οκτωβρίου 2009 σε 21 κράτη-μέλη. Και σε αυτή την γνωμοδότηση αναφέρεται στις, στα κενά όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων υποστήριξη των σιδηροδρομικών, της εφαρμογή των μέτρων του σιδηροδρομικού πακέτου. Αναφερθήκα στο σημείο 2, κατάλογο κρατών μελών. Πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός διότι δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη τον ίδιο βαθμό σοβαρότητας ως... και ούτε τις ίδιες ελλείψεις. Λάβετε τα αυτό υπόψη. Αν θέλετε να δακτυλοδείξετε κάποιον θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι δεν έχουν όλα τα ίδια κράτη-μέλη την ίδια κατάσταση. Εντοπίστηκαν κενά όσον αφορά τρία βασικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα έλλειψη ανεξαρτησίας των χειριστών των υποδομών όσον αφορά τους σιδηροδρόμους, ανεπαρκή εφαρμογή μέτρων της οδηγίας για, την, για τα τέλη που καταβάλλω την πρόσβαση στις ιδρομικές γραμμές, διότι δεν πληρώνονται, δεν συμπεριλαμβάνονται στο άμεσο κόστο των συνδρομικών υπηρεσιών. Υπάρχει έλλειψη κινήτρων για τον διαχειριστή των υποδομών να μειώσει το κόστο και τα τέλη. Τα κράτη-μέλη δεν ισορροπούν τον προπολογισμό των χειριστών των υποδομών και υπάρχει έλλειψη ε, ελέγχου των διαφόρων σχημάτων επιδόσεων και επίσης δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι ρυθμιστικοί φορείς με τι αναγκαίε εξουσίες να διορθώσουν προβλήματα ανταγωνισμού στον τομέα των σιδηροδρόμων. Αυτά αντικατοπτρίζουν ότι σε κάποιες χώρες σίγουρα υπάρχει μια τάση προστασίας των ιστορικών επιχειρήσεων των συνδρομικών από τον ανταγωνισμό, διότι το πακέτο ήθελε να σαγάγει πλήρη ανταγωνισμό και να ανοίξει την αγορά των σιδηροδρόμων τίνεται να κατηγορείται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καθυστερημένη δράση κατά αυτών των κενών, για την κάλυψη των κενών. Αυτό κατά την άποψή μου αποτελεί μία απλούστευση. Α, αυτό που αναφέρεται στη σημεία 3 και 5 λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρά σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από τη συνθήκη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι κοινοποιούνται όλες οι, όλα τα εθνικά μέσα που υπάρχουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να ξεκινήσει ξεκίνησε τον Απρίλιο 2003 διαδικασία παράβασης κατά όλων των κρατών μελών, διότι δεν κοινοποίησαν εθνικά μέτρα. Το 2003 δεν υπήρξε καμία κοινοποίηση για την εκείνη τη διαδικασία. Για τα νέα η εφαρμογή ε, ξεκίνησε από το Μάιο 2004 οι 10 κράτη-μέλη και τον Ιανουάριο 2007 για Ρουμανία και Βουλγαρία, δηλαδή τη στιγμή της προσχώρησης. Ε, η οδηγία επίσης επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υποβολή εκθέσεω σχετικά με την εκτέλεση που εκδόθηκε τον Μάιο του 2006 και βασιζόταν σε λεπτομερή μελέτη της αγοράς των σιδηροδρόμων και αυτό ήταν ένα κρίσιμο βήμα διότι η έκθεση εμπεριέχει κριτήρια που εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάλυση των διευρωπαϊκών δικτύων σχετικά με την ανάλυση της εφαρμογής του νόμου από τα κράτη-μέλη. Χωρίς αυτά τα κριτήρια θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προσφύγουμε κατά των κρατών μελών. Ήταν η βάση για τον έλεγχο της εκτελέσεως και εφαρμογής του νόμου που ξεκίνησε τότε μετά το 2006 και το 2007 στείλαμε δύο γύρους ερωτηματολογίων σε 25 κράτη-μέλη. Αυτό το πακέτο εμπειρία είχε πάρα πολλές διατάξεις εφαρμοστικές και τα κράτη-μέλη, όπως γνωρίζετε, έχουν το δικαίωμα να στέλνουν όλα τα έγγραφα στις εθνικές τους γλώσσες. Οπότε υποχρεωθήκαμε να κάνουμε μετάφραση όλων αυτών των εγγράφων και αυτό χρειάστηκε χρόνο. Πέραν αυτού, οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπάθησαν να επιφέρουν συμμόρφωση με συγκριτικό τρόπο με τα κράτη-μέλη, δηλαδή χρειάστηκαν πολλές συνεδριάσεις, πάρα πολλές συζητήσεις και πολλές επαφές. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στόχος ήταν να προκαλέσουμε αλλαγή και όχι απλώ να κατηγορούμε και να στρεφόμαστε με επιχειρήματα κατά κρατών μελών. Αφού λάβαμε, λάβανε, λάβαμε τα ερωτηματολόγια, στείλαμε 24 επιστολές, επίσημες κοινοποίησεις στα κράτη-μέρη τον Ιούνιο του 2008, πήραμε τις απαντήσεις, γίνανε και άλλες συνεδριάσεις και τώρα είμαστε στη φάση στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε την, γνωμοδότηση τον Οκτώβριο, την αιτιολογημένη γνωμοδότηση τον Οκτώβριο του 2009. Κατά την άποψή μα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τα μέσα που διαθέτει και συμφωνούμε ότι η πλήρης εφαρμογή του πακέτου για τους σιδηροδρόμους είναι μια προϋπόθεση για την άνοιγμα των αγορών στο σιδηροδρομικό τομέα, διότι το πακέτο δημιουργεί τις αναγκαίες θεσμικές συνθήκες χωρίς τις οποίες το άνοιγμα της αγοράς δεν θα λάβει χώρα και θα καθυστερήσει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη-μέλη αρνούνται να εφαρμόσουν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα έχει επιλογή παρά τα κράτη-μέλη αυτά να τα στείλει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να προσφύγει κατά αυτό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πριν σας δώσω το λόγο, να επανέθω σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα που ετέθη από τον κύριο Κούν, θυμάμαι καλά, για την παροχή υπηρεσιών για το τι συνέβη τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά θα μπορούσαν να βρεθούν στην έκθεση για την αγορά των σιδηροδρόμων που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Αναφέρετε την έκθεση αυτή στο ψήφισμά σας. Υπήρχε συγκεκριμένο ερώτημα που ετέθη από την κυρία Γιάλα Σέντερ για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε από κάποια εταιρεία σιδηροδρομική που ζήτησε πρόσβαση στην αγορά σε γειτονική χώρα, από ό,τι γνωρίζουμε, έγινε αίτηση για παραχώρηση δυναμικού, αλλά δεν ακολουθήθηκε από αίτημα χορηγήσεως πιστοποιητικού, άρα δεν υπήρξε απόρριψη πρόσβαση στην αγορά, αλλά δεν διεκπαιρεώθηκε η διαδικασία. Επίσης, ετέθη ερώτημα από κύριο Μπιλμπάου γιατί τα κράτη-μέλη δεν εφάρμοσαν ε, τα μέτρα του πακέτου. Έχουμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα που δημοσιεύτηκε και για κάθε κράτος μέλος λεπτομερώς αναφέρουμε τα κενά και τις ελλείψεις. Αυτό το υπόμνημα θα μπορούσε να διατεθεί σε όλους σας για να καταλάβετε καλύτερα την κατάσταση. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρχουν ισότιμες συνθήκες για όλους και γι' αυτό η αναφορά που κάνατε κάποιοι στην ανάγκη να παρασχεθούν επαρκείς υποδομές είναι μια πρόταση που μοιραζόμαστε και επίσης η πρόταση σχετικά με τη δημιουργία ισότιμων συνθήκων που πρέπει να επικρατούν όσον αφορά τις εξωτερικές πτυχές των μεταφορών. Με άλλα λόγια, εσωτερήκευση εξωτερικών δαπανών, όχι μόνο για το σιδηροδρόμους, αλλά και για άλλες μορφές μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ με σεβασμό προς τον κύριο Στέρξ που ακολουθεί η έκθεσή του. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, συνοψίζοντας και απαντώντας τα όσα υπόθηκαν. Άκουσα αυτά που είπατε και προσβλέπω στις τροπολογίες σας και αν θέλετε να ενισχύσετε το κείμενο με τα χαράς να το κάνω διότι είναι δικό σας ψήφισμα, απλώς έχει το όνομά μου μετά χαράς να το κάνω αυτό. Ισχύουν πολλά από αυτά που άκουσα όσον αφορά τις επενδύσεις κυρίως για τις υποδομές και το καθεξής. Εγώ πάντα θεωρούσα, κύριε Καστελέτη, ότι όταν ένα δημόσιο υπάλληλο πήγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρώτο που έπρεπε να κάνει θα ήταν να πάει σε μια μικρή αίθουσα και του βάζανε ένα τσιπάκι πίσω από το αυτί του που λέγανε απελευθέρωση των αγορών, ενιαία αγορά είναι ο Θεός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, κάποιος σας αφαίρεσε το τσιπάκι όσον αφορά τους σιδηροδρόμους και πραγματικά το λέω με κάθε ειλικρίνεια, μακάρι να είχαμε δει τέτοιο ζήλο που είδαμε στην απελευθέρωση της ενέργειας, την απελευθέρωση της πολιτικής αεροπορίας, απελευθέρωση όλων των άλλων τομέων, ταχυδρομικών υπηρεσιών. Μακάρι να είχαμε δει τέτοιο ζήλο που είδαμε σε αυτούς τους τομείς που παρουσιάστηκε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να το βλέπαμε για τους σιδηροδρόμους. Πραγματικά είναι πρόβλημα μεγάλο για μας. Δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί καταφέραμε να ακολουθήσουμε το δρόμο της ενιαίας αγοράς στην απελευθέρωση σε τόσους άλλους τομείς, αλλά στους ιδηλοδρόμους αποτύχαμε. Και ο λόγος για τον οποίο αποτύχαμε, κατά την άποψή μου, είναι διότι υπήρξε έλλειψη συντονισμένης προσπάθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για να ε, πετύχουμε αυτήν την αγορά και γι' αυτό σας κατηγορούμε και ίσως θα πείτε ε, βεβαίως κάνουμε ό,τι μπορούμε και κάνουμε αυτό και εκείνο και μπορείτε να το υπεραπλουστεύσετε και δεν μπορείτε να το εξετάσετε σε επίπεδο 100 μελών και μπορώ να σας βρω άλλους 9 λόγους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παρότι γιατί κάναμε. Και αν το κάνουμε αυτό, πέφτουμε στην παγίδα σιδηροδρόμου. Στην Βουδαπέστη την περσμένη εβδομάδα και άκουσα του ουγγρικού σιδηροδρόμου που, που ξεκίνησαν τη συζήτηση λέγοντα Χρειαζόμαστε παρέκκληση από το πρώτο πακέτο σιδηροδρόμου. Ξεκίνησαν τη συζήτηση έτσι. Και βεβαίω ε, έμειναν ε, ε, εμβρόντιτοι, δεν καταλάβαναν ότι ήμουν στην αίθουσα και σε απάντηση του είπα να τα πάλι, οι Ουγγρικοί σιδηρόδρομοι δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα που μαστίζει τους σιδηροδρόμους και εδώ μιλάει σιδηροδρομικός, έτσι. Εγώ αγαπώ τους σιδηροδρόμους μου που σας μιλάω. Και εδώ έχουμε την απογοήτευση. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση σε αυτό το κοινοβούλιο για την έλλειψη δράσης σε αυτό το τομέα. Υπάρχει καχυποψία, να το πω ειλικρινά. Είμαστε καχύποπτοι. Πιστεύουμε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν κινηθήκατε είναι γιατί φοβόσαστε το Συμβούλιο. Αυτή είναι η υποψία. Μπορεί να κουνά τα κεφάλι του τα μέλη, περισσότεροι γνέφουν. Άλλοι κουνά το κεφάλι, περισσότεροι ναι, γνέφουν. Λοιπόν, έκλεισα αυτό. Παραμένει γεγονός. Το 2001, 15 κράτη-μέλη προσυπόγραψαν αυτό το πακέτο των σιδηροδρόμων. Όταν τα νέα κράτη υπέγραψαν την συνθήκη προσχώρησης και αυτές οι χώρες υπέγραψαν αυτό το πακέτο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες, αλλά αυτό που βλέπω στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι ότι η δικαιολογία του πρώτου πακέτου σιδηροδρόμων ή τα προβλήματα του πρώτου σιδηροδρομικού πακέτου μετακυλίεται ως δικαιολογία για το ότι δεν συμβαίνει τίποτα όσον αφορά τους, ε, τις επενδύσεις στους σιδηροδρόμους τους. Τα προβλήματα των Ουγγρικών σιδηροδρόμων, τα προβλήματα των Βαλτικών χωρών, τα προβλήματα της Ρουμανίας ε, ε ισχύαν πολύ πριν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλλειψη επενδύσεων, έλλειψη δέσμευσης ε, της κυβέρνησης να υποστηρίξει ο δρόμος σε κάποιες από τις χώρες που δεν αναφέρεται και που εφαρμόζει τα μέτρα ε, είναι η Φιλανδία που έχει εύρος ε, μεταξύ σιδηροτροχιών αντίστοιχο με τη Ρωσία. Άρα το πρόβλημα αποστάσεων σιδηροτροχιών δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι θέμα διελειτουργικότητας. Δεν θα έπρεπε να σταματά την εφαρμογή ε, του πρώτου πακέτου των σιδηροδρόμων. Τέλος πάντων, όπως έλεγα, ε, θέλω να δω τι θα μου δώσετε σαν προτάσει, τροπολογίες, Για να προχωρήσουμε, αυτό που φαίνεται ότι είναι ηλίου φαϊνότερο είναι ότι αυτή η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει ότι αυτό το πρώτο πακέτο των συνδρόμων θα εφαρμοστεί από όλα τα κράτη-μέλη. Προτιμούμε βέβαια, κύριε Καστελέτη, θα προτιμούσαμε κατά τη διάρκεια της δικής μας ζωής. Σας εύχομαι μακρόν βίων, φωνάζει ένας βουλευτής. Να σας πω για τα τυπικά. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών η 5η Μαΐου. Προθεσμία για τροπολογίες 5 Μαΐου, ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών 1 Ιουνίου, Ολομέλεια Ιουνίου. 5 Μαΐου λοιπόν η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. 5 Μαΐου. Θα με ρωτούσατε ίσως, έλεγα θα με ρωτήσετε ποια χρονιά, ε. 5 Μαΐου 2010. Κύριε Στέρξ, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Η έκθεσή σας όσον αφορά τις διαδικασίες για τα σκάφη και πού βρισκόμαστε. Ευχαριστώ. Ξέρετε ότι προσπάθησα ε, Ja, dus dat ik nog bezig ben op vraag van het Spaanse voorzitterschap om te proberen. Μου ζήτησε η Ισπανική Προεδρία να καταφέρουμε να πετύχουμε σε πρώτη ανάγνωση. Μετά από διάφορες συναντήσεις με την Προεδρία πάντως, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει να προχωρήσουμε πολύ. Δεν ξέρω ποιος πρέπει να προτείνει το συμβιβασμό. Αλλά δεν ξέρω αν θα λυθεί το ζήτημα. Είμαστε στην ηλεκτρονική επικοινωνία αλλά πιστεύω ότι δεν είναι για τα τελωνία και Υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα για ηλεκτρονική επεξεργασία. Το Συμβούλιο πάντως πέντε χρόνια προσπαθεί να καταλήξει κάπου. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα σκάφη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην υποφέρουν από τις διατυπώσεις, αλλά για θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης κτλ. Εγώ συμφωνώ, αλλά το Συμβούλιο ζητά διάφορες παρεκκλήσεις για άλλα πράγματα με τα οποία εγώ δεν συμφωνώ. Την ημερομηνία πρέπει να την κρατήσουμε. Συμφωνούμε μία γλώσσα. Για τα υπόλοιπα υπάρχουν διάφορα μικρά πράγματα που δεν μας απασχολούν. Τώρα την επόμενη εβδομάδα θα συγκεντρώσω τους σκιώδεις συζητητές για να τους ενημερώσω. Έχω ετοιμάσει κάτι γραπτά για την τελευταία συνεδρίαση. Να έχουμε κάτι ώστε μεταξύ σκιωδών να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα συναντηθώ και με την Προεδρία και για μένα είναι στόχος να πετύχουμε ε, στην πρώτη ανάγνωση. Καλό θα ήταν αυτό. Είναι ε, αισιόδοξο βέβαια, έχοντας δει την ημερήσια διάταξη του Μαΐου που είναι η έκθεση και απάνω, μου φαίνεται όμως υπερβολικά αισιόδοξο. Γι' αυτό μήπως να πάμε τον Ιούνιο στην Ολομέλεια Αλλιώς δεν βλέπω πώς θα τα καταφέρουμε αν πρέπει να περιμένουμε και τις μεταφράσεις, να έχουμε συζητήσει με τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Δεν νομίζω να προλαβαίνουμε. Πάντως, σε πρώτη ανάγνωση, εγώ θέλω να πετύχουμε συμφωνία. Αλλά σίγουρα δεν θα πρέπει να κάνουμε πολλές υποχωρήσεις εμείς στο Κοινοβούλιο ή τέλο πάντων δικιά μας Επιτροπή. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Στέρξ, λέει ο Πρόεδρος, πριν πάρουν το λόγο σκιώδης εισηγητές. Τότε θα έλεγα να προχωρήσετε στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, ώστε να είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό να το κάνετε. Κύριε Κούν. Και εγώ ευχαριστώ τον κύριο Στέρξ ε, για αυτή την έκθεση. Και ο κύριος Στέρξ ε, ε, είναι εμπειρογνώμονα σε ό,τι αφορά ζητήματα ναυτιλιακά και η επικοινωνία μας ε, είναι πολύ καλή. Ε, ο κοινό ε, στόχος σε ό,τι αφορά την δημιουργία ενό τέτοιου ενιαίου χώρου χωρί σύνορα στην Ευρώπη είναι, έχει ήδη ξεκινήσει δηλαδή να, να καταστούν και οι μετακινήσεις μικρών αποστάσεων ελκυστικές και οικονομικά βιώσιμες αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει βέβαια να λαμβάνονται υπόψη και οι κανόνες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Πράγμα το οποίο θέλουμε και, δεν θέλουμε και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Δεν θέλουμε δηλαδή να ισχύουν διαφορετικά πράγματα στην Ευρώπη και διαφορετικά όταν θα είμαστε στο παγκόσμιο επίπεδο διεθνή παίκτη. Ε, πράγματι, ε, σε ό,τι αφορά την αλλαγή πληροφοριών θα πρέπει αυτό να ισχύσει γενικά, ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών, έτσι καλλιώς ε, τα ηλεκτρονικά ημερολόγια σκάφους έχουν ήδη ε, ξεκινήσει να τηρούνται ε, και εδώ καλύπτεται και ο τομέας της αλληλείας, όχι μόνο των μεταφορών και κάτι τέτοιο βέβαια σε τελική ανάλυση οδηγεί σε μεγαλύτερη ασφάλεια στις θάλασσες. Εκείνο όμως το οποίο επιθυμούμε είναι η κυκλοφορία των σκαφών τα οποία μετακινούνται μόνο ανάμεσα στου λιμένε των κρατών μελών, που ελέγχονται δηλαδή τελωνιακά Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ορισμένε παρεκκλήσει για αυτό το είδος κυκλοφορίας, ώστε να μην υπάρχουν, να μην παρεμποδίζονται ειδικότερα για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τα κανονικά δρομολόγια ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς λιμένες ε, ε, σε ό,τι αφορά ορισμένες υποχρεώσεις, σε ό,τι αφορά το προσωπικό πλοίαρχο, πλοίαρχος, ε, πολύ συχνά ο οποίος μεταβαίνει κάθε εβδομάδα και εκτελεί αυτό το δρομολόγιο, γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό το δρομολόγιο και δεν χρειάζεται κάποιος επιπρόσθετος επόπτης για αυτή την περίπτωση, ο πάλι, όπως λέγεται. Αυτά και ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά για την εκθέσή σας. Μιλάνα. Ο Μιλάνα. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Στέρξ, περισσότερα κομπλιμέντα από αυτά που έκανε ο πρόεδρος ε, πριν. Πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Αυτή του κυρίου Στέρξ εργαστήκαμε σοβαρότατα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσει την εντολή του αυτή για μεσολάβηση και σε επαφές με το Συμβούλιο. Επαναλαμβάνω αυτό που είπε ο κύριος Στέρξ και τα είπαμε κατηδίαν. Το θέμα της γλώσσας είναι σημαντικό να παραμείνει σαν θέμα ε, διαφοροποίηση μεσοπρόθεσμα της εφαρμογής του μέτρου. Συμφωνώ, μεν, να παραμείνει το 2013 σαν ημερομηνία εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων, όμως αφορά τη γλώσσα, για να θα μπορούσαμε να καθυστερήσουμε κατά δύο-πέντε χρόνια για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα, αλλά θα πρέπει να παγιωθεί η αρχή. Θα ήμουν αντίθετο να διαφοροποιήσουμε τους λιμένες και ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα μικρό λιμάνι μπορεί να έχει παρέκκληση όσον αφορά τη γλώσσα. Αυτό θα σήμαινε περιπλοκή την ζωή των λιμένων, δηλαδή να κάνουμε το αντίθετο από αυτό που θέλουμε να κάνουμε. στο μεγάλο λιμάνι είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιηθούν τα αγγλικά από ότι σε ένα μικρό λιμάνι πιθανότατα. Θα επέμενα προς αυτή την κατεύθυνση όσον αφορά την εφαρμογή, αυστηρή εφαρμογή το 2013, ελπίζοντας ότι με στεναρότητα θα αντιμετωπίσετε το Συμβούλιο. Υπάρχει ομοφωνία γύρω από τη θέση σου και θα ήταν χρήσιμο να προχωρήσει μέχρι τέρμα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα συνδέονται με το πώς θα προχωρήσει και θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία των διαπραγματεύσεων και που θα καταλήξει. Ευχαριστώ κυρία Φώστερ. Λοιπόν, πριν από την ακυρωθήσα ουσιαστικά ολομέλεια του Στρασβούργου της περασμένης εβδομάδας, το συζητήσαμε, σε υποστηρίξαμε ένθερμα. Το ξέρεις, κάποιοι είχαμε κάποιες διαφορές όσον αφορά την προθεσμία εφαρμογής. Ε, διαφορά δύο ετών. Ε, δεν ήταν τίποτα σοβαρό σαν πρόβλημα για τις ομάδες. Πραγματικά προσπαθήσαμε όλοι μαζί να το κάνουμε να πετύχει. Όσον αφορά το που βρίσκεσαι τώρα, όπως είπες, φαίνεται σαν να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο σε κάποιους από τους τομείς. Έχεις πολύ καλή εντολή που σου δώσει η Επιτροπή αυτή, να πας εκεί πέρα, να προβάλλεις τα επιχειρήματά σου, προφανώς αυτό έκανες, αλλά να τα ενισχύσεις, να το τονώσεις τα επιχειρήματά σου, γιατί εδώ βρισκόμαστε. Όπως σου είπα η ομάδα μας, υποστήριξε το 2015 σαν εναρκτήρια ημερομηνία και πολλοί άλλοι υποστήριξαν το 2013. όπω σου είπα, κοίτα, σου λέω, πρέπει να καταλήξουμε συμφωνία. Θα είμαστε ευέλικτοι στο ECR για αυτό το θέμα. Αν μπορεί να πετύχει το 2013, καλώς. Ίσως να θέλουν να το πάνε στο 2014, αλλά έχεις την υποστήριξή μας αν μπορείς να πας το 2013, γιατί θέλουμε να προσπαθήσουμε να επιληθεί το θέμα αυτό, όπως καταφέραμε να λύσουμε τα προβλήματα στην πρώτη ανάγνωση. Όσον αφορά αυτό που είπες για την χρήση χαρτιού κλπ. Ε, δεν είμαι τόσο σίγουρη, το αφήνω σε σένα το πώς ασχολούνται τα λιμάνια με αυτό. Ε, ε, το θέμα είναι ότι αυτοί θα πρέπει να κάνουν κάτι. Δεν θέλουμε ένα μικρό λιμάνι να κλείσει, μικρή επιχείρηση να κλείσει. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας στην Επιτροπή αυτή. Αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε. Όμως κάτι τελευταίο όσον αφορά το γλωσσικό, ένα από τα ισχυρότερα προβλήματα. Ίσως να μπει σε αιτιολογική σκέψη αντί για άρθρο, αυτό ζητήθηκε, ε, αναφέρθηκε αυτό. Το θέμα των γλωσσών. Ποιο ήταν το πρόβλημα. Είναι θέμα ασφάλειας. Όσο αμφιβολίες μπορείς να βγάλεις από την επικοινωνία, κυρίως στις θαλάσσιες μεταφορές, από, από τους διάφορες μορφές μεταφορών, τόσο σε καλύτερη θέση είσαι. Δεν είμαστε αντίθετοι όσον αφορά τα μικρά λιμάνια ή χώρους πολύ περιορισμένους που δεν χρειάζεται να κάνεις διδακτορικό στα αγγλικά για να δουλέψεις σε πλοίο αλλά είχαμε επιχειρήματα γιατί θα πρέπει ε, να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση όπως κάναμε επί σειρά δεκαετιών και στις αερομεταφορές. Θα πρέπει να επιμείνεις στη θέση σου. Πού θα πρέπει να μπει αναφορά, θα πρέπει να είναι σε άρθρο η αναφορά αυτή στη γλώσσα. Μπορεί να τεθεί χρονοδιάγραμμα, κάποια παρέκκληση λογική για να εφαρμοστεί, αλλά εμείς είχαμε λόγους για τους οποίους θέλαμε να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Όπως σας είπα, από τη δική μας άποψη, Έχεις πλήρη υποστήριξη της ομάδας μας και σου ευχόμαστε καλή τύχη όταν πας ξανά να τους ξαναδείς. Ο κύριος Γκράντες Δε Πασκουάλ, σκιώδης του ΕΛΚ. Ζητώ συγγνώμη, γιατί επειδή στην αρχή δεν υπήρχε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη, είχα μπερδευτεί. Μετά μου είπαν ότι έρχεται η έκθεση του κυρίου Στέρξ και έτρεξα. Εν πάση περιπτώσει, Κύριε Στέρκ, δεν θα κουραστώ ποτέ να πω καλά λόγια για τη δουλειά σας. Το ίδιο και σε αυτή την περίπτωση και για τις διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Μπράβο. Εδώ στην αρχή ήμουν πολύ σκεπτικός για το τι είναι εφικτό και τι δεν είναι. Η ίδια η Ισπανική Προεδρία θέλει το θέμα αυτό να κλείσει σε πρώτη ανάγνωση, να εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση. Και έτσι από την αρχή εγώ είδα ότι ήταν θέματα που θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Δεν είναι θέμα ισπανικό εξάλλου, ούτε και το γλωσσικό. Έτσι λοιπόν, Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, δεν είναι τόσο σοβαρό Μιλήσαμε σήμερα και για τις αεροπορικές μεταφορές και τα μέτρα που ισχύουν, αλλά βλέπετε στη θάλασσα δεν υπάρχει αυτή η συνένεση για απλοποίηση των πάντων και να κρατήσουμε τα αγγλικά σαν γλώσσα επικοινωνίας χωρίς να χρησιμοποιούμε άλλες γλώσσες. Ίσως το πρόβλημα εδώ, και μπορεί να μην θέλει να το δεχτεί ο εισηγητής, είναι να λάβουμε υπόψη μας σε μια αιτιολογική σκέψη ίσως και όχι σε ένα άρθρο, έναν τέτοιο προβληματισμό. Πολλές φορές λέμε ότι το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Δεν αξίζει τον κόπο να κάνουμε λοιπόν την προσπάθεια. Γιατί οι διαφορές που υπάρχουν σε αυτή την έκθεση δεν είναι τόσο μεγάλες. Είναι εξαίρετη κατά τα άλλα. Οπότε θα ήθελα ο συγκητής να κάνει μια προσπάθεια αυτές τις διαφορές να τις αμβλύνει και ως σκιώδης θα ζητούσα να βοηθήσουμε προσπαθώντας να πετύχουμε μια συμφωνία με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Καραμίτσος, φίλος μας είναι. Οπότε μην τον στριμώξετε πολύ και ο Καραμίτσος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι ελπίζω να είμαστε καλοί φίλοι. Έχουμε μακρά ιστορία συνεργασίας. Μέσω πακέτων είτε όχι μέσω πακέτων. Είναι δυνατόν να συνεργαστούμε με τον εισηγητή για να καταλήξουμε συμφωνία ταχύτερο δυνατόν. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα καταφέρουμε προ την πρώτη ανάγνωση. Δεν ξέρω η Ισπανική Προεδρία έδωσε κάποια προτεραιότητα. σω τα καταφέρουμε λοιπόν. Πράγματι υπάρχουν δύο-τρία προβλήματα που εκκρεμούν. Θα ήθελα να προσθέσω και άλλο ένα και ζητώ συγγνώμη. Όσον αφορά το, την ηλεκτρονική και την ε, μορφή τη χάρτινη, όσον αφορά τη γλώσσα. Το πρόβλημα τη γλώσσα μπορεί να επιληθεί αν ακολουθήσουμε την ηλεκτρονική προσέγγιση στο τέλο και ξεχάσουμε το χαρτί διότι τα... είναι τυποποιημένα τα έντυπα, οι φράσει είναι τυποποιημένε. Ακόμα και ένα Ρώσο καπετάνιο που δεν μιλάει άλλη γλώσσα παρά τη ρωσική μπορεί να πατήσει να κλικάρει στο συγκεκριμένο σημείο και το μήνυμα να περάσει στα αγγλικά μέσω ηλεκτρονική μορφή στο safety net ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Μπορούμε να βρούμε κάποια λύση, πιστεύω. Από την άλλη, πράγματι, στην πρακτική, στι θαλάσσιε μεταφορέ, όπω οι αερομεταφορέ αυτέ τι μέρε, τουλάχιστον τι μέρε μα, τουλάχιστον στι περισσότερε περιπτώσει, χρησιμοποιούνται τα αγγλικά. Είναι κάτι τυποποιημένο. Ήδη υπάρχει σύμβαση που απαιτεί εκείνου που είναι στο κατάστρωμα να μιλάνε ε, αγγλικά. Στο χώρο διακυβέρνηση του σκάφου, μάλλον στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται στα μεγάλα σκάφη. Στα μικρά σκάφη όμως δεν ισχύει αυτό. Δεν βλέπω όλοι να, που μεταφέρουν πράγματα μεταξύ των ελληνικών νησιών και της ε, Ελλάδα Ελλάδας να μιλάνε αγγλικά. Τις περισσότερες φορές το κάνουν γιατί μιλάνε αγγλικά για άλλους δικούς τους λόγους, για τουριστικούς λόγους Φερρυπίν. Αλλά ε, εκεί είναι η διαφορά. Το άλλο είναι ο χρονισμός. 2013 είναι ενδεχόμενη ημερομηνία διότι και το Safe θα είναι έτοιμο από την πλευρά μας, σύμφωνα το πακέτο του πακέτου και το e-customs θα υπάρχει. Ε, λίγοι μήνες παραπάνω μπορούν να δοθούν σαν συμβιβασμός ίσως. Θα ακολουθήσω την πρόταση της κυρίας Φώστερ. Ίσως λίγους μήνες μπορούμε να δώσουμε. Μη σκοτωνόμαστε και όλα, μπορούμε να πετύχουμε συμβιβασμό και κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω προς τον εισηγητή εφόσον θα συζητά το θέμα με την Προεδρία. Μια μικρή μας ανησυχία θέλω να εκφράσω έχουμε αυτή τη γενική προσέγγιση για τις εκχωρηθήσεις ε, πράξεις, ε, για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Ε, λέγαμε συνήθως έχουμε πέντε χρόνια μετά πάμε για συναπόφαση. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αυτό που έχουμε στο παράρτημα είναι ένας κατάλογος. Δεν εμπεριέχει τίποτα παραπάνω από έναν κατάλογο σημείων που είτε είχαμε στη συναπόφαση πριν ή μορφές ε, μέτρων του IMO που θα επεκταθούν. Δεν είναι κάτι ουσιαστικό που λέμε ότι αν ε, προσθεθεί άλλο είδους ε, φάκελος ή οτιδήποτε επικοινωνία χρειάζεται απόφαση συμβουλίου. Ε, χρειάζεται συναπόφαση. Το Συμβούλιο μας είπε δίνουμε πενταετία και μετά πάμε στην απόφαση. Είναι πολύ σκληρό, πολύ διοικητικό, εκεί θα έπρεπε να υπάρχει αυτόματη παράταση, διότι αυτού του είδους η οδηγία που έχουμε είναι απλούστατη ε, είναι κάτι που πρέπει να το εξηγήσουμε περισσότερο στο Συμβούλιο. Γιατί δεν έχει νόημα να εφαρμόζεται αυτό εδώ, να εφαρμόσουμε εδώ αυτό που εφαρμόζουμε σε, άλλους πιο περίπλοκα, σε άλλα πιο περίπλοκα τεχνικής φύσεως παραρτήματα. Εδώ είναι πιο απλά τα πράγματα. Ε, αυτό ήθελα να πω. Δεν χρειάζεται να επανέλθουμε πάνω σε αυτό μετά από μια πενταετία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Κύριε Στέρξ, θέλετε να συνοψίσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ του συναδέλφου και φυσικά θα είμαστε σε επαφή ώστε μέχρι τον Ιούνιο να έχουμε τελειώσει με το κείμενο. Είναι πολύ σημαντικό. Κάθε αναβολή είναι μειονέκτημα. Είναι σε βάρος μας. Ελαστικότητα όσον αφορά τη γλώσσα και όπως λέει και ο κύριος Καραμίτσος, υπάρχουν διεθνείς κανόνες και μπορούμε να προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε. Στην πράξη θα δούμε. Ακόμα και εδώ στην Επιτροπή μας ε, η πλειοψηφία ήταν μικρή. Οπότε θα δούμε και αυτό. Για την ημερομηνία. Θα δούμε, είναι μάλλον εύκολο. Αλλά δεν θα πω ότι ό,τι υπάρχει για την υποχρέωση κάποιας δήλωσης ή αναγγελίας που έχει να κάνει με τις μεταφορές, εντάξει, αλλά όχι με τα τελωνία, όχι με θέματα υγείας κλπ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε το σύνολο. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα όπου όλα τα στοιχεία εκεί μέσα που πρέπει να βασίζονται σε κάποια χαρτιά να συμπεριλαμβάνουν ό,τι πρέπει. Ο κύριο Τεγκράντε που λέει ότι μπορεί μια χώρα να ζητήσει παρέκκληση, αν πρόκειται για υγεία, για μετανάστευση κλπ. Το δεχόμαστε. Αλλά υπάρχουν πράγματα, κείμενα, για τα οποία δεν συμφωνώ, γιατί διαλύουν το σύστημα. Εσείς είπατε ότι εφόσον υπάρχει ένα πρόβλημα με την ασφάλεια, με τη μετανάστευση, με την υγεία, ένα κράτος να μπορεί να πει ότι δεν δίνω μια πληροφορία αν μπει ένα σκάφο, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα λόγο και να λέει το κράτο ότι έχω ένα λόγο που το ζητάω αυτό και γι' αυτό το ζητάω. Τότε ναι. Αλλά να πούμε ότι θα ισχύει μόνο για τι μεταφορέ και όχι μόνο για τα τελωνία κλπ. Όχι. Δεν συμφωνώ. Πρέπει να είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, ένα πλήρε σύστημα και να πούμε ότι αυτό το σύστημα πρέπει να παραμείνει έτσι ολόκληρο. Με ενιαία θηρίδα για όλους όσους εμπλέκονται. Είμαστε πολύ κοντά στο σωστό αποτέλεσμα και η Επιτροπή ελπίζω να έχει κείμενο στην επόμενη συνεδρίαση. Άμα έχουμε το κείμενο θα έχουμε τέσσερις κολόνες, τέσσερις στήλε και εκεί θα είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό με στην επόμενη εβδομάδα ήταν δυνατόν να το φροντίσει η Επιτροπή. Άκουσα πάντως τις παρατηρήσεις σας, άκουσα τι ζητάτε να είμαστε και αυστηροί αλλά και ελαστικοί για να πετύχουμε συμφωνία και ότι η Προεδρία επίσης είναι πρόθυμη να προχωρήσει για να έχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Πρέπει να αποφεληθούμε από αυτή την θετική διάθεση. Ευχαριστώ πολύ και τους συναδέρφους και εσάς Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Στέλξ. Έχετε την εντολή από εμά να συνεχίσετε τις διαπραγματεύσεις σας. Και σας ευχαριστώ και για την υπομονή που επιδείξατε μέχρι να φτάσουμε στην εκθεσή σας. Τελειώσαμε λοιπόν μέχρι τις 3 σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ.